Μάλιστα. Ελπίζω όλοι να βρήκατε τις θέσεις σας. Και η επόμενη... το επόμενο πάνελ θα πραγματευτεί τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους άτομα με αναπηρία 2020-2030 καθώς και ένας ε, συνεκτικός ε, Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτό είναι το αντικείμενο της, του επόμενου πάνελ και έχω πάρα πολλούς ε, ομιλητές μαζί με την ε, κυρία Κούντα Άνκα, τη συμπρόεδρο, μέλος ε, του EDF, της Εκκληστικής Επιτροπής του Φόρουμ για τα τόμα με αναπηρία. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας πω δύο λόγια για την έκθεση η οποία εγκρίθηκε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, την προηγούμενη εβδομάδα, με συντριπτική μάλιστα πλειοψηφία. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή στρατηγική σε ό,τι αφορά την αναπηρία. Μια, ένα έγγραφο, μια έκθεση πολύ σημαντική για όλους σας. Τα διάφορα λοιπόν θέματα, 8 στον αριθμό, αποτέλεσαν τις 8 προτεραιότητες μας σε ό,τι αφορά θέματα ε, προσβασιμότητας, συμπερίληψης, ισότητας, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κοινωνικής προστασίας, υγείας και εξωτερικών σχέσεων σε ό,τι αφορά τις επαφές μας και με τρίτες χώρες. Αυτές ήταν οι οκτώ κορυφαίες προτεραιότητές μας, λοιπόν. Και η έκθεση ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη συνειδητά επιλέξαμε να συγγράψουμε την έκθεση αυτή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρία για, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους τυφλούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κοφούς καθώς και με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία για τον αυτισμό και την Mental Health Europe, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ψυχική Υγεία. Ε, περιλαμβάνονται λοιπόν πολλοί παράμετροι, πολλές παράμετροι στην έκθεση αυτή συμμετείχαν και τα μέλη των εθνικών αντιπροσωπιών. Η έκθεση λοιπόν καταρτίστηκε από κοινού με εσάς και χάρη στις δικές σας ε, παρατηρήσεις και σχόλια έχει πάρει τη μορφή που έχει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταφέραμε να φτάσουμε σε πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα έγγραφο εργασία. Δεν είναι έγγραφο το οποίο θα καταλήξει κάπου σε ένα σιρτάρι στον πάτο κανένα Θέλουμε να δώσουμε μήνυμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κρατημέλη προκειμένου να κινητοποιηθούν εδώ σε ό,τι αφορά την ισότητα των ευκαιριών, σε ό,τι αφορά την ισότητα των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Γιατί διαπιστώνουμε ότι πολλά άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια. Εμπόδια τα οποία δεν ε, καταλύονται. Και η έκθεση λοιπόν ε, ζητά από εσά να προβείτε σε συστάσεις σε προτάσεις για βελτίωση της καθημερινής σας ζωής. Σας χρειαζόμαστε λοιπόν. Οι αρχές σας είναι αυτές στις οποίες θα πρέπει να αποταθείτε και να τους πείτε, κοιτάξτε, αυτή η έκθεση εδώ έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άτομα με αναπηρία και περιλαμβάνει πολύ καλές προτάσεις. Εσείς είστε αυτοί που θα πρέπει να κάνετε το λόμπι για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Γιατί αν παραμείνει σε επίπεδο εγγράφου, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Κυρία Επίτροπε, κυρία Τέισεν, ελπίζω και εσείς ε, να θέλετε να κάνουμε τη διαφορά μαζί μας. Ε. Μίλησα πολύ ώρα όμως και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Άνκα. Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας αγαπητοί συναδελφοί. Φίλοι, σας καλωσορίζω όλους ε, σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή. Όλοι σας έχετε έρθει για να μιλήσουμε θέματα τα οποία είναι τόσο ουσιώδη για όλους μας άτομο αναπηρία. Και μου αρέσει πραγματικά αυτή η φράση που άκουσα του κυρίου Ταγιάννη σήμερα το πρωί. Είπε ότι μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες και την ελευθερία αλλά παράλληλα μιλάμε και για συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου αυτές οι τόσο σημαντικές για μας αξίες να καταστούν πραγματικότητα. Να καταστούν πραγματικότητα όχι μόνο για κάποιους από εμά, αλλά για όλους μας. Για όλους όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως εκ τούτου σήμερα, εδώ, στη συζήτηση αυτή για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία. Θέλουμε όλα τα μέρη που συμμετέχουν να συνέλθουν. Έχουμε εκπροσώπους από την πολιτική ζωή, από τα συνδικάτα. Έχουμε επίσης εκπροσώπους και των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία. Και πιστεύω ότι πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κινούμαστε από τα όμορφα λόγια στα συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις οι συγκεκριμένες πράξεις αυτές οι οποίες μπορεί να γίνουν αισθητές όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάπου στις Βρυξέλλες, αλλά συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα γίνουν αισθητές και ορατές και απτές στα εθνικά κράτη-μέλη. Εδώ στο Βέλγιο, σε ένα, σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε εμά, στη Λετωνία, από όπου και είμαι. Οι συνθήκε, συνθήκες, ένας διαστρωμένο διάλογος στον οποίο κάθε οργάνωση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για Ευρωπαϊκή, Περιφερειακή, Εθνική Ένωση και Οργάνωση, θα μπορούσε να συμμετάσχει προκειμένου να αλλάξουμε τις πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα και τα... αυτά που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Μόνο μια τέτοια προσπάθεια θα καταστήσει τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία θα λάβει σαρκα όχι να παραμείνει στο επίπεδο της υπογραφής, της επικύρωσης, να μπει σε ένα ράφι κι αυτή. Όχι, να καταστεί πραγματικότητα. Και να δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να ζήσει μια ανεξάρτητη ζωή ως μέλος της κοινωνίας, ανεξάρτητα από το που ζει ο καθένας. Και ε, μιας και δεν έχουμε χρόνο για μακροσκελές εισαγωγές, να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις στο πάνελ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Άνκα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαία Επίτροπο, κυρία Μαριάν Τέισεν. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδροι, μάλλον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλοί μου φίλοι. Είμαι, Είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι εδώ στο τέταρτο Ευρωκοινοβούλιο των ατόμων με αναπηρία. Αυτό είναι το αποκορύφωμα μιας ε, ε, εορταστικής χρονιάς και για την Ευρώπη και για το Ευρωπαϊκό Αναπηρικό Κίνημα. Πριν από ένα ακριβώς χρόνο γιορτάσαμε την δέκατη επέτειο της ε, υιοθέτησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ήταν μια στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας και αίσθησης ε, μεγάλου κατορθώματος, γιατί ήταν η πρώτη φορά που μία σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, οντότητα. Και μάλιστα μετά από τόσα χρόνια ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και με τη συμπερίληψη πριν από 20 χρόνια της πάταξης των διακρίσεων στις ιδρυτικές συνθήκες. Επίσης, πριν από 20 χρόνια ιδρύθηκε και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ατόμων με αναπηρία και θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι το EDF γιατί χάρη σε εσά η φωνή των ατόμων με αναπηρία, των ανδρών και των γυναικών ακούγεται ηχηρά και στεντόρια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόλις την περασμένη Πέμπτη εκφώνησα ομιλία στην ε, συζήτηση στην Ολομέλεια που σας ανέφερε η Χέλγα με θέμα την πρόοδο σε ό,τι φορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία για την περίοδο 2020-2030. Και είπα ότι μέχρι το 2020 ένας στους πέντε Ευρωπαίους υπολογίζεται ότι θα έχει κάποια αναπηρία. Και είπα ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν είναι να γινόμαστε όλο και πιο μικροί, αλλά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα εφαρμόσουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και μετά το 2020. Πιστεύω ότι η σημερινή διάσκεψη ε, μας δίνει ήδη μια εξαιρετική ευκαιρία για να το κάνουμε. Και μάλιστα μια κοινωνική δικαιοσύνη και μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην μένει κανείς πίσω. Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίε, έχουμε αναλάβει τουλάχιστον τρει δεσμεύσει που καθοδηγούν τις δράσεις μας. Καταρχήν, αποκοινούμε τα κράτη-μέλη. Έχουμε τη νομική υποχρέωση να, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη συμβατή με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, όλα τα ε, θεσμικά όργανα ε, ανακήρυξαν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του κοινωνικού εταίρου. Αυτό ο πυλώνας είναι μια ισχυρή δέσμευση υπέρ των δικαιωμάτων όλων, υπέρ τη ίση μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών, που φυσικά συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα αυτά και τα άτομα με αναπηρίε. Και τρίτον, προσυπογράφουμε τους βιώσιμους στόχους ε, της ανάπτυξης και των Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα βιώσιμους ε, αναπτυξιακούς στόχους για όλους ε, και φυσικά και για τα άτομα με αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική των Ατόμων με Αναπηρία μας καθοδηγεί κατά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και τον περασμένο Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε μια διεξοδική έκθεση προόδου. Κάτι που δείχνει ότι τα άτομα με αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το συνολικό επίπεδο ανεργίας, απασχόλησης μάλλον, συγγνώμη, είναι 71%. Ενώ για, τους, για τα άτομα με αναπηρία το επίπεδο απασχόλησης είναι 48%. Μόνο 27% των ατόμων με αναπηρία έχουν αποφοιτήσει από τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και ένας στους τρεις ανθρώπους με αναπηρία διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Θα πρέπει να διορθώσουμε τις, ε, τις αδικίες αυτές, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Χρειαζόμαστε και τα δικά σας ταλέντα και το δικό σας δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευτυχώς γίνει πιο προσβάσιμη ε, και το διαδίκτυο είναι πιο προσβάσιμο, ιδιαίτερα οι ιστοσελίδες των δημόσιων φορέων. Επίσης, ε, προσυπογράψαμε και η ένταξή μας στη συνθήκη του Μαρακές θα κάνει περισσότερα δημοσιεύματα και βιβλία προσβάσιμα. Ενισχύσαμε και τις διατάξεις προσβασιμότητας στα δημόσια έργα, στις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές και στις σχετικές νομοθεσίες. Και ελπίζω ότι του χρόνου θα υιοθετήσουμε επιτέλους και τη δική μου πρόταση για μια ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη περί προσβασιμότητας. Και στην αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών θα υπενθυμίσω στους υπουργούς την υποχρέωση που έχουν να κάνουν πραγματικότητα αυτή τη νομοθετική πράξη. Κάπου αλλού που πραγματικά επιφέρουμε διαφορές είναι η ελεύθερη διακίνηση με την οδηγία για, την, για τις υπηρεσίες υγείας, το πιλωτικό πρόγραμμα για την κάρτα του ατόμου με αναπηρία που θα αξιολογήσουμε του χρόνου, με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τους κανόνες συντονισμού για τα μακροπρόθεσμα υγειονομικά επιδόματα και επίσης το, η ενίσχυση του προγράμματος Erasmus με το έρασμο ΣΥΝ. Αυτά είναι μερικά μόνο λίγα παραδείγματα που αποδεικνύουν εμπράκτο την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών δράσεων. Βέβαια πολλά έχουμε ακόμη μπροστά μας, πολλά θα πρέπει να υλοποιήσουμε στο μέλλον. Θα πρέπει ήδη να σκεφτούμε από τώρα τους μελλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία. Θα λάβουμε υπόψη και τις τα, τα τελικά συμπεράσματα της Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη και το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της περασμένης εβδομάδας που σας εξήγησε η κυρία Χέλγα Στίβενς. Και επίσης ε, θα εισακουστεί και η δική σας συμφωνία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και για να χρησιμοποιήσω και το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία, Τίποτα για σας χωρίς εσάς. Η δική σας φωνή πρέπει να ακουστεί σε αυτή τη συζήτηση. Θα οργανώσουμε λοιπόν δημόσιες διαβουλεύσεις για να έχουμε άμεσες πληροφορίες απευθείας από εσά. Και στην πρώτη συζήτηση που έχει ε, προγραμματιστεί για, τον, για την άνοιξη του 2018 για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού. θέλουμε και τη δική σας συνεισφορά. Θα πρέπει να προλιάνουμε το έδαφος για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου ε, να γίνει μια ε, αξιόλογη ε, εξέταση του τι έχει γίνει μέχρι τώρα και μία αντίληψη για το ποιες προσκλήσεις απομένουν μπροστά μας. Και το, ένα πολύ σημαντικό θέμα, ο προϋπολογισμός. Πάνω από 268.000 άτομα με αναπηρία έχουν επωφεληθεί από δραστηριότητε που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία συμβάλλουν και στην ανάπτυξη των ε, θεμελιωδών στοιχειωδών υπηρεσιών για μια ανεξάρτητη διαβίωση. Και στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανεξάρτητη διαβίωση που θα υιοθετήσει το Συμβούλιο Υπουργών αύριο. Και φυσικά οι συζητήσεις ε, για τα οικονομικά είναι περίπλοκες. Πολλό δε μάλλον σήμερα από το πιθανό αντίκτυπο που θα έχει και το Brexit στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα, τα ταμεία μας μετά το 2020 δεν θα πρέπει να δαπανούν, να μην κόβουν ούτε ένα ευρώ για τα άτομα με αναπηρία. Θέλω να βελτιώνουμε το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας. Θέλω ένα προϋπολογισμό που θα επενδύει σε δυναμικό που θα στηρίζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα, τον Πυλώνα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα είναι συμβατός με, την Ευρωπαϊκή, με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Και ελπίζω σε αυτό να με υποστηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα κλειδί να πω ότι μόνο από κοινού θα καταρρίψουμε τους φραγμούς και τα εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ήρθα εδώ για να ακούσω εσά ε, του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στη συζήτηση και αυτοί ήρθαν να ακούσουν εσάς. Γι' αυτό περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ. Yeah. Ε, ευχαριστώ. Ε, αντιπρόεδρος του, της Ευρωπαϊκής Διακομματικής Ομάδας ε, για τις ε, αναπηρίες. Η κυρία Χαρκίνη, σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας κυρίε και κύριοι. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω που ήρθατε, σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ σήμερα, γιατί μας δίνει αυτό μια ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας και πιο σημαντικό να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Γιατί κάτι που ξέρω στα σίγουρα είναι ότι όσοι δεν έχουμε αναπηρία, όσοι δεν έχουμε έναν στενό συγγενή με αναπηρία, δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνει το να ζει με αναπηρία κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και αυτό το μάθημα το έμαθα μόνο πρόσφατα, να σας πω την αλήθεια. Και ντρέπαμε που σας λέω παρά το γεγονός ότι είμαι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Διακομματικής Ομάδας για τα άτομα με αναπηρία, μόλις ε, για πρώτη φορά φέτος ε, είχα και προσέλαβα έναν υπάλληλο, μία υπάλληλο, μία νεαρή γυναίκα με αναπηρία και μόνο όταν ε, προσλάβαμε αυτή τη νεαρή γυναίκα καταλάβαμε τι ακριβώς σημαίνει. Το Airbnb που νίκιαζε διαφήμιζε ότι είναι προσβάσιμο. Δεν ήταν όμως η πραγματικότητα όπως προέκυψε. Και να σας πω ότι αν δεν βοηθούσαν οι υπόλοιποι βοηθοί μου τη γυναίκα αυτή να δουλέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα τα κατάφερνε. Αυτή η νεαρή λοιπόν γυναίκα μας έφερε και μας δίδαξε ένα πολύ πολύτιμο μάθημα και σε μένα και στους υπόλοιπους βοηθούς μας. Και χαίρομαι που βρισκόμαστε στην ίδια πλατφόρμα και με την Επίτροπο, η οποία έχει καταθέσει σημαντικέ και πολύ καλέ προτάσει και με την κυρία Χέλκα Στίβεν, η οποία πρόσφατα κατέρτισε μια εξαιρετική στρατηγική για την αναπηρία. Όλοι μα λοιπόν τα κάνουμε αυτά, αλλά σε κάποιο βαθμό είμαστε σε απόσταση. Μόνο όταν εκτίθεται κανεί και έχει πραγματικέ εμπειρίε από πρώτο χέρι καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό ακριβώ. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και να σας θερήσω το χρόνο μιλώντας για νομοθεσία, γιατί νομίζω ότι θα έχετε ακούσει λίγο πολύ τι γίνεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Δεν θέλω όμως να υποτιμήσουμε και τη σημασία της ε, ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στην νομοθεσία. Έχουμε και τη σύμβαση του ΟΗΕ, η οποία όμως ε, αν η νομοθεσία δεν είναι γνωστή και την υποτιμούμε, είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι κενή ε, περιεχομένου. Θέλω να μιλήσω για δύο πράγματα. Καταρχά, ω αντιπρόεδρο τη ε, διακομματική ομάδα για την αναπηρία, και να σα δώσω μόνο ένα-δύο στοιχεία, σαν παράδειγμα, για το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και στο επίπεδο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το EDF, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, που μας δίνει υποστήριξη και αρρωγή και πολλά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Διακομματική Ομάδα μας. Δίνει λοιπόν πολλά, πολλές πληροφορίες και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και πιστεύω ότι είναι πραγματικά α, πολύτιμη η συμβολή τους. Αλλά στην παρούσα φάση, στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, είναι η εφαρμογή της ε, συνθήκης ε, της, του ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε μαζί μας... Ε, πολίτες ε, και συναδέλφους από όλη την Ευρώπη. Ελπίζω να μην σας πειράξει το γεγονός ότι σήμερα θα αναφέρω την Ιρλανδία συγκεκριμένα, η οποία είναι μία από τις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση του ΟΗΕ. Και θα ήθελα να να την ευκαιρία αυτή, να καλέσω την Ιρλανδία να επικυρώσει εδώ και τώρα την ε, Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ. Όλοι όμως ασφαλώς γνωρίζουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο η επικύρωση, το θέμα είναι η υλοποίηση. Και πρόσφατα, τα τελευταία δύο χρόνια, λάβαμε τις, ε, τα τελικά πορίσματα για το πώς τα πηγαίνουμε εμείς εδώ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και από εκεί και πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάστηκε στενά για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι θα έχει πραγματικό νόημα και δεν θα είναι κενά λόγια. Είναι ιστορική αυτή η στιγμή ότι πρόκειται δηλαδή για την πρώτη φορά που ένα σώμα ανθρώπινων δικαιωμάτων προέβησε σε υποβολή συστάσεων προς το Κοινοβούλιο. Και τώρα, όπως σας είπα, δουλειά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα αυτό το πακέτο συστάσεων. Περιλαμβάνει και μεγάλες λεπτομέρειες. Ε, για παράδειγμα, ο προπολογισμό, τα χρονοδιαγράμματα, η εποπτεία δεν είναι κάτι το οποίο απλά το γράφουμε και το ξεχνάμε. Όχι, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε όλα αυτά. Ε, μερικοί άλλοι στόχοι τώρα. Οι ιδέε τι οποίε περιλαμβάνουμε στη δουλειά μα στην διακομματική ομάδα, είναι η εξασφάλιση τη ελεύθερη κυκλοφορία. Όλοι οι υπόλοιποι, ξέρετε, θεωρούμε την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένη, αλλά για άτομα με, με αναπηρία θέματα όπω η προσβασιμότητα, η βοηθών είναι κρίσιμη σημασία. Κάτι που μπορούμε να κάνουμε ως Κοινοβούλιο είναι να εξασφαλίσουμε ότι κάποια από τα προγράμματά μας, για παράδειγμα, το Εράσμους, στην παρούσα φάση συζητάμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα λοιπόν αυτά θα είναι προσβάσιμα για νέους ε, όταν ε, περνάνε σύνορα. Δύο άλλα θέματα περιλαμβάνουν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ή αλλιώς προπολογισμό. Την τελευταία φορά Αυτή τη φορά μάλλον θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα μας τα προγράμματα, όλες μας οι πολιτικές και το καθεξής θα έχουν λάβει υπόψη τη διάσταση της αναπηρίας. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε στον επόμενο προϋπολογισμό. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία μας απασχόλησαν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ε, ανεκτές, προσβάσιμες τις συνεδριάσεις μας, κάποιες συνεδριάσεις μας ε, στο κοινό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Helga Stevens γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετική η βοήθειά της και μας έμαθε πάρα πολλά. Τελευταίο σχόλιο. Στις 12 το πρωί σήμερα, μαζί με την Evelyn Κεπχαρτή, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και υπεύθυνη για θέματα IT, παραβρεθήκαμε στην ε, προβολή μιας ταινίας η οποία είχε δημιουργηθεί από το προσωπικό IT του Κοινοβουλίου και μας έδειξαν τις προσπάθειες που καταβάλουν οι ίδιοι υπάλληλοι για να εξασφαλίσουν ψηφιακή προσβασιμότητα για τους συναδέλφους τους. Και ξέρετε κάτι, είναι σημαντικά αυτά συνάδελφοι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι με αναπηρία είναι κάπου αλλού, αλλά είναι συνάδελφοι, γιατί κάτι που ξεχνάμε διαρκώς είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να καταστεί σε οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του. Και το προσωπικό του τμήματο αυτού του Κοινοβουλίου έχει εργαστεί άκοπα και σκληρά για το σύστημα αυτό το οποίο είναι σημαντικό για τους συναδέλφους τους και πραγματικά αποτελούν υπόδειγμα για όλους μας. Θεωρώ ότι όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να κάτσουν να δουν αυτό το φιλμ. Δεν είναι αρκετό να καταρτήσουμε νομοθεσία. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Και η ταινία κλείνει με ένα ερώτημα. Τι θα γίνει με εσά, εσύ, τι μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι το ερώτημα που όλοι καλόμαστε να απαντήσουμε. Ευχαριστώ, συναδέλφα Χάρκιν. Μία μικρή αλλαγή θα ήθελα να κάνουμε στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όλους σας κατά πόσον το σύστημα με τους υποτίτλους λειτουργεί ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να διαβάσει τους υποτίτλους από τη θέση του, από το έδρανο του, θα μπορούσαμε να φροντίσουμε να μεταφερθεί πιο κοντά στην οθόνη. Να το πείτε στους κλητήρες παρακαλώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βαρδακαστάνη. Έχει κάποια ανακοίνωση να μας κάνει και νομίζω ότι σίγουρα θα ξέρει καλύτερα τι θέλει να σας πει από εγώ. Thank you. Ευχαριστώ, ο ε, κύριος Βαρδακαστάνης. Τέλειο Οκτωβρίου του 2015 που η επίτροπο που κάθεται στα δεξιά μου ήρθε στην εκτελεστική επιτροπή που συνεδρίαζε τότε εδώ στι Βρυξέλλε και συναντηθήκαμε για περίπου μία ώρα κράτησε αυτή η συνεδρία. Είχαμε να συζητήσουμε το κείμενο για την προσβασιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα δημοσιοποιείται και αυτό γίνεται φέτος 2 12 του 2015 τήρησαν την υπόσχεσή τους και της Κομισιόν είπα δε εγώ ότι τόσα χρόνια που δουλεύω στα θεσμικά όργανα δεν θυμάμαι κανέναν άλλο επίτροπο να τηρεί τόσο πιστά την υπόσχεσή του. Οπότε ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Το Σεπτέμβριο φέτος το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ανέκρινε μια κοινή θέση που αφορά αυτήν την πράξη για την προσβασιμότητα. Αύριο δε, όπως ήδη μας είπε η Επίτροπος, ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο πρόκειται να εγκρίνει μια τέτοια γενική κοινή θέση. Και σήμερα θα εγκριθεί το σχετικό ψήφισμα. Οπότε και αμελητή να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια το Συμβούλιο. Όσο αφορά αυτή την κοινή ε, θέση για την πράξη που αφορά την προσβασιμότητα. Πριν όμως να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα, αυτό το κείμενο, θέλω να πω το εξή. Κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε μαζί σας ότι χρειάζεται κάποια στρατηγική στεγανή για την προσβασιμότητα για την περίοδο 2020-2030 ούτω ώστε να υλοποιηθεί η σύμβαση του ΟΗΕ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να σας βοηθήσουμε προς το και πριν το τέλος της εντολής σας, ούτω ώστε να μείνει κάποια σχετική πρόταση για την επόμενη επιτροπή. Αλλιώς θα χάσουμε χρόνια, εάν πρόκειται να διτυπώσει την πρόταση για επόμενη επιτροπή. Κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να εορταστεί η δεκάτη επέτειος της ε, σύναψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, Σύμβασης στη συνέχεια της συνολής του 2001. Παρακαλούμε να επιληφθείτε. Και δεν το λέω αυτό για λόγους τελετουργικούς. Είναι σημαντικό την αρχή της δεκαετίας που ξεπροβάλλει θα πρέπει τα κέντρα που βάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ε, οι ίδιοι τώρα στις απαρχές της νέας στρατηγικής της ελπιζόμενης καινούργια εποχής να μπορούμε να αφήσουμε αυτό το αποτύπωμα, το θετικό, αυτό το κληροδότημα σε σχέση με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει προσβασιμότητα όχι μόνο από πλευράς υποδομών, ίντερνετ κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα όσον αφορά τα δικαιώματα και να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους οι πολίτες. Και τώρα, συνάδελφοι συμφωνείτε αύριο να απευθυνθούμε στο Συμβούλιο να μην καθυστερεί άλλο. Καλώς και σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Χέλγα. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε τον κύριο Βαρτακαστάνη. Είναι σαφές το μήνυμα το οποίο μεταφέρετε και θα ήθελα να συνεχίσω με το πρόγραμμα και τους ομιλητές. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Θα σας ζητήσω λοιπόν να τηρήσετε τα χρονικά όρια, γιατί αλλιώς το θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος στην αίθουσα να πάρει το λόγο. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Μιλιο Ράιλι. Η διαμεσολαβητής. Thank you Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, αξιότιμοι καλεσμένοι κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω του διοργανωτέ που με προσκάλεσαν σε αυτή τη βαρισίμαντη εκδήλωση, μια και είμαι μέλο τη ε, Επιτροπή ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που παρακολουθεί την εφαρμογή τη Σύμβαση του ΟΗΕ. Το τελευταίο Ευρωκοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρία έγινε το 2012 αμέσω μετά την κύρωση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η αρχή μιας πολλά υποσχόμενης αλλά πολύ δύσκολης πρωτοβουλίας ε, να ε, βάλουμε σάρκα και οστά σε μια σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και μάλιστα κατάλαβα πολύ καλά ω Ιρλανδοί πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία, γιατί όπω είπε πριν από λίγο η Μάριαν, η Ιρλανδία είναι το τελευταίο κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ακόμη κυρώσει την σύμβαση. Κάτι που με θλίβει ιδιαίτερω. Ελπίζω να ληφθούν υπόψη αυτές οι σημαντικές κατευθυντήρες γραμμές που δίνει η Επιτροπή και μάλιστα μια πραγματική προσήλωση του θέματος των ατόμων με αναπηρία σημαίνει μεταφέρουμε τα λόγια ε, που βρίσκονται στη θεωρία σε απτούς ε, τρόπους που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε πτυχή του της καθημερινότητάς τους και να γίνουν σεβαστά αυτά τα δικαιώματα. Ο Ευρωπαίος ε, Μεσολαβητής ε, δέχεται κυρίως παράπονα και καταγγελίες. Και μάλιστα οι καταγγελίες που αφορούν ε, άτομα με αναπηρία καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα. Προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών κτηρίων, παιδιά με αναπηρία και έχουν πρόβλημα με τα, την επιστροφή ιατρικών εξόδων, χρήση της διαμηνίας τη νοηματική που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετοχή στι στις διαγωνισμούς Μάλιστα, τα συμπεράσματα της ειδική αυτής επιτροπής ε, εμπνέουν το στρατηγικό μου έργο στον τομέα αυτό. Και θα σας δώσω μερικά από τα παραδείγματα. Το 2016, μετά τις παρατηρήσεις της Αρμόδιας Επιτροπής και την υποβολή σχετικών καταγγελιών, ξεκίνησα μια στρατηγική έρευνα για το κατά πόσο η αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία από το Κοινό Καθεστώς Υγειονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το JSIS, είναι συμβατό με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. Η πλήρη αποζημίωση των ιατρικών εξόδων από το κοινό αυτό καθεστώ υγειονομική ασφάλιση προβλέπεται, αλλά μόνο για σοβαρή νόσο. Για να θεωρηθεί όμω μία νόσο σοβαρή, θα πρέπει να πληρούνται τέσσερα κριτήρια. Και ένα από αυτά είναι ε, το μειωμένο προσδόκιμο ζωής είπα στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούγκερ, ότι αυτή η ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας δεν ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση του κοινωνικού μοντέλου που προωθεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Πολλές αναπηρίες δεν περιορίζουν αναγκαστικά το προσδόκιμο ζωής. Παρ' όλα αυτά έχουν τεράστιο κόστος και ιατροφαρμακευτικό και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματική και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Ξεκίνησα λοιπόν στοχευμένες διαβουλεύσεις ε, με ενώσεις ε, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναπηρία ή που κάποιο συγγενή του έχει αναπηρία, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Και μάλιστα για κάποιε προτάσει του. Ε, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει αν κάποιες διατάξεις ε, του κοινού καθεστώτος υγειονομικής ασφάλισης θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να γίνουν συμβατές με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Επίσης, να υιοθετηθεί ένας ε, ενδεικτικός κατάλογος ε, ιατροτεχνολογικών προϊόντων που θα τύχουν πλήρους επιστροφής εξόδων και αυτό θα πρέπει συζητάτε με εκπροσώπους των αναπηρικών οργανώσεων και υπαλλήλων των της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς εφαρμόζεται εμπράκτος το, κοινωνικό καθεστώς, το κοινό καθεστώς υγειονομικής ασφάλειας και κατά πόσο εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Μας ενδιαφέρει επίσης η προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Πέρυσι χαιρετήσαμε την υιοθέτηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των δημόσιων φορέων. Και παρόλο που αυτό δεν ισχύει για τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογέ για τα κινητά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παροτρύνονται να τηρήσουν αυτέ τι απαιτήσει προσβασιμότητα. Μάλιστα, τον Ιούλιο ξεκίνησε μια στρατηγική έρευνα για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων τη Κομισιόν και των online μέσων. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποσχέθηκε ένα πιλωτικό σχέδιο για επιλεγμένες σελίδες ε, μιας διοργανικής πύλης του ίντερνετ προκειμένου να ε, προσφέρει ευανάγνωστες ε, πληροφορίες και κάποια ε, μαθήματα υποχρεωτικά προσβασιμότητας για το προσωπικό. Και μάλιστα το εφαρμόζουμε αυτό και στις υπηρεσίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που έχουμε μεταφρασμένες 24 γλώσσες τα στοιχεία μας και ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της προσβασιμότητας. Έχουμε ένα επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ. Μάλιστα πρόσφατα έχουμε υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με το ιστοσελίδα για τα θέματα αυτά. Ε, μία σημαντική πρόκληση θα είναι να ε, εφαρμόσουμε, να υλοποιήσουμε τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Και είναι σημαντικό αυτό. Φυσικά το χρονοδιάγραμμα, η παρακολούθηση και η σαφήνεια είναι πολύ σημαντικά. Πρόσφατα παρακολούθησα ένα πρόγραμμα στην ε, Βρετανική τηλεόραση που παρακολουθεί τι προσπάθειε 10 ατόμων με αναπηρία στην ε, αναζήτηση μιας θέση εργασία. Και μάλιστα με ε, τράβηξε την προσοχή μου μία γυναίκα που έχει προβλήματα κινητικότητας λόγω κεφαλικής παράλυσης και προσπαθεί να βρει θέση δημοσιογράφου. Και μάλιστα χρειάστηκε τρεις ώρες με, δημόσιες, με δημόσια συγκοινωνία για να πάει από το σπίτι της ε, στο χώρο εργασίας, ε, σε μια προσωρινή θέση της απασχόλησης που της, που προσφέρθηκε. Και μάλιστα δεν καταδέχτηκε να πει στους συναδέλφους της πόσο ταλαιπωρήθηκε και πόσο πονούσε για να μην ε, την, τη λυπηθούν. Πραγματικά τέτοια, ε, τέτοιος άνθρωπος όπως και, άλλοι, και άλλα άτομα με παρόμοια προβλήματα δεν θα πρέπει να φοβούνται ε, ότι θα αντιμετωπιστούν με διακρίσεις. Ήρθε η στιγμή να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταπεξέλθει στις ε, προσδοκίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποτελέσει παράδειγμα προ μίμηση στον τομέα τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Eh, Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Οράιλη. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει ως διαμεσολαβήτρια και ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω την κατανόηση για τη διάφορα, αν θέλετε, της προσέγγισης της ιατρικής και της προσέγγισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο ασθενείς. Ε. Όσο πιο πολύ το κατανοήσουν αυτό, τόσο πιο καλή θα είναι η κατανόηση του θέματος. Ε. Και τώρα το επόμενο άτομο που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριο ε, Λούκα Βισεντίνη, Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το φόρουμ για να εκπροσωπήσω εδώ την Συνομοσπονδία Συνδικάτων τη Ευρώπη ε, και να συμμετάσχουμε σε αυτή την σημαντική συζήτηση με εντυπωσίαση εισοδόρμη εδώ σε αυτή η αίθουσα γιατί ποτέ ξέρετε δεν έχω δει αυτή την αίθουσα, αυτό το μικύκλιο γεμάτο όπως εσείς το γεμίσατε σήμερα οπότε συγχαρητήρια capacity, ε, to... μπράβο, μπράβο που μπορέσατε να κινητοποιήσετε όλους αυτούς, αυτούς όλους τους ανθρώπους να βρίσκονται εδώ για αυτή τη σημαντική σημερινή συζήτηση. Το δεύτερο τρόπο που θέλω να σας πω έχει πιο προσωπικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Ιταλική αντιπροσωπεία των ατόμων με αναπηρία. Αυτή που σήμερα είναι κοντά μας πρόκειται για φίλους. Έχω συνεργαστεί μαζί τους στο παρελθόν όταν ήμουν συνδικαλιστή στην ε, χώρα μου. Θα ήθελα λοιπόν να τους απευθύνω αυτόν τον προσωπικό θερμό χαιρετισμό. Πρέπει έχουμε τώρα στα αγγλικά. Τι είναι ε, η ETUC, η συνομοσπονδία μας. Έχουμε ε, 19 ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες μάλλον. Προσβούμε 45 εκατομμύρια εργαζομένων και από αυτούς πολλοί έχουν αναπηρία. Άρα Είμαστε σύμμαχοι εκπροσωπεί ένα τον άλλο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι στρατηγικέ μας είναι συντονισμένε έτσι θα αποσπάσουμε καλύτερα αποτελέσματα για αυτούς που και εσείς και εμείς εκπροσωπούμε σήμερα. Να επισύρω την προσοχή σας ε, στα όσα προτάσουν τα συνδικάτα μας ούτω ώστε να ενσωματωθούν, να ενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά τα πρόσωπα με αναπηρία. Φυσικά θα πρέπει ε, να εξασφαλιστεί το ότι θα σεβαστά τα σχετικά δικαιώματα, ιδίω στην αγορά εργασία για αυτούς που προσπαθούν να μπουν στην ε, αγορά απασχόληση, αλλά δεν μπορούν γιατί υπάρχουν διάφοροι φραγμοί και δυσμενείς ε, διακρίσεις. Και επίση σημεία προσανατολισμού είναι για εμάς η σύμβαση του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο πολύ σημαντικό. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και πρόσφατα έχουμε το θεματολόγιο του ΟΗΕ για το 2030 για τους βιώσιμους στόχους, τους αναπτυξιακούς. Και επίσης η συμφωνία του Γκέτεμπορ, τόσο πρόσφατη. Να σας πω για ακριβώς αυτόν τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης. Θεωρούμε ότι πρόκειται για επίτευγμα γιατί ξαναγυρίζει ε, στην προβληματική για αυτή η υπόθεση γιατί πρόσφατα ε, ξεχάσαμε λόγω της λιτότητας τα κοινωνικά μας πρότυπα, το κοινωνικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Σχεδόν το γκρεμίσαμε άρα να επανέλθουμε σε αυτές τις κοινωνικές αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων είναι μια αρχή και αφορά και την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες που δικαιούνται βοήθειας, υποστήριξης να ζήσουν με αξιοπρέπεια κάποιων υπηρεσιών για να συμμετάξουν στην αγορά απασχόληση στην κοινωνία σε ένα περιβάλλον εργασιακό σύμφωνο με τις ανάγκες τους. Αξιοπρέπεια επομένω και ενσωμάτωση. Κοινέ ανάγκες, δικαιώματα όσων έχουν αναπηρίες, αλλά αυτά αφορούν και κάθε άλλο Ευρωπαίο, κάθε Ευρωπαίο εργαζόμενο και στην Ευρώπη και παντού σε όλο τον κόσμο. Άρα είναι κοινό μας συμφέρον επίτευξη αυτών των στόχων και να το πετύχουμε θα πρέπει να μπει φρένο στην λιτότητα σε αυτές τις περικοπές των συστημάτων πρόνοιας και δημοσίων παροχών και υπηρεσιών. Διαφορετικό μείγμα πολιτικής χρειάζεται για επενδύσεις ιδιωτικής και δημόσιας, αλληλεγγύη, και σύγκληση προς τα πάνω. Θα πρέπει όλες οι αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα να ενσωματωθούν σε κάθε ευρωπαϊκή πολιτική, ιδίω στις συνθήκες, αλλά και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια στον κοινωνικό προπολογισμό για αυτές τις αρχές του κοινωνικού πυλώνα και έτσι να βοηθηθούν αυτοί που έχουν αναπηρέσει επίση να υπάρξει ξεκάθαρο χάρτη πορεία για αυτήν την υλοποίηση. Ένα πρόγραμμα δράση να τα συμφωνήσει το Συμβούλιο και να τα υλοποιήσει κάθε κράτο μέλο. Τι εννοούμε όμω με αυτό. Εννοούμε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη έχετε αναφέρει τις νομοθετικές πληροφορίες ε, και επίσης συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η ζωή του κόσμου. Να σας αναφέρω όσον αφορά τους εργαζομένους κάποια παραδείγματα. Η αρχή της ενσωμάτωσης όσων έχουν αναπηρίες, αλλά και όλες οι άλλες αρχές του κοινωνικού πυλώνα. Και έτσι να έχουμε πραγματικά μία απασχόληση που ενσωματώνει την κοινωνία και κανείς δεν μένει πίσω. Ίση μεταχείριση για απασχόληση, για εργασία. Οι υλοποίηση στα κρατημέλη θα πρέπει να εποπτεύεται, να είναι πιο αποτελεσματική. Η πρόσβαση στην ε, εργασία με συγκεκριμένα μέτρα από την πρόσληψη θα πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στα ταλέντα της δεξιότητας όσων έχουν ε, αναπηρία. Όλες εκεί εργασιακέ συνθήκε, να είναι προσαρμοσμένε στα όσα πρέπει και να υπάρχει ισότητα, εγγυήσει προ τούτο για ισότητα όσον αφορά την αμοιβή, την ισορροπία ιδιωτικού με δημοτικού βίου και να απαγορεύεται, να υπάρχει αποτροπή από οποιαδήποτε είδου δυσμενή διάκριση. Αλλά τα πρόσωπα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες για σταδιοδρομία, ακριβώς όπως έχουν και όλοι οι εργαζόμενοι. Είναι στόχοι που θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να εφαρμόσουν με συλλογική διαπραγμάτευση αλλά και νομοθετικά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει βέβαια δυσανάλογο βάρος για τους εργοδότες, γιατί το θα αποτελεί κάποια πρόφαση να προβούν σε μία εφαρμογή, σε κάποιο είδους ε, διακρίσεις. Να μην έχουμε κοινικό διαχωρισμό, να μην πέφτουν στην φτώχεια οι άνθρωποι με αναπηρία, θα πρέπει να φροντίσουμε επομένως την προσβασιμότητα στην απασχόληση και θα πρέπει η γενιά μας να χειραφετήσει τους νέους, να πιάσουν τόπο οι ικανότητές τους. Απασχολησιμότητα, ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία παιδεία, κατάρτιση για τις δεξιότητες, εξέλιξη προσωπική, στοχευμένη. Πριν κανείς μπει στην αγορά απασχόλησης, πριν κανείς πιάσει δουλειά να μπορεί, ακόμα και αν χάσει τη δουλειά του, να ξαναμπεί στην αγορά εργασία. Να μην περιθωριοποιούνται οι άνθρωποι μια αναπηρία μέσω της ανεργίας και η κοινωνική πρόνοια θα πρέπει να φροντίζει για την ένταξη όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να δούμε τις ανάγκες τους για κάθε απασχόληση και να υπάρχουν κάποιες ε, διατάξεις που θρακίζουν και προστατεύουν αυτούς που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Επόμενος προσβασιμότητα σε όλους, προστασία, υποστήριξη σε αυτούς που έχουν αναπηρία και τις οικογένειές τους. Αυτά είναι οι στόχοι μας. Η κοινή, σας διαβεβαίω, ότι τα συνδικάτα είναι στο πλευρό σας για την επίτευξη αυτών των στόχων και όπως προείπα τα συνδικάτα και οι συνεργατικές οργανώσεις θα πρέπει οι δικές οργανώσεις να είναι σύμμαχοι για προστασία και ενσωμάτωσή σας. Θα πρέπει μαζί να χτίσουμε μια κοινωνική Ευρώπη που όπως ανέκαθεν λέει ο πρώτος Γιούνκερ, μια Ευρώπη που προστατεύει. Πιστεύω μαζί θα το πετύχουμε και σας ευχαριστώ. Dank Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βυζεντίνη, για την παρουσίασή σας. Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα. Θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην επόμενη αμολήτρια, την κυρία Hainsworth. Έχετε το λόγο. Και παρακαλώ να τηρήσετε το χρονικό όριο. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σήμερα το απόγευμα στο 4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα άτομα με αναπηρία. Ονομάζομαι Τζάνα Χέινσουαρθ και είμαι εκλεγμένη πρόεδρο τη κοινωνική πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα που συνενώνει 47 ευρωπαϊκά δίκτυα κοινωνία των πολιτών και ενώσεων τη κοινωνία των πολιτών. Τα μέλη μα είναι ενωμένα στην αποστολή να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια για όλου. Να προωθήσουν την κοινωνική συμπερίληψη και την εξάλληψη τη φτώχεια και για να προωθήσουν το δικαίωμα όλων στην κοινωνία να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Διάφορα από τα μέλη μας ε, εργάζονται κυρίως ό,τι αφορά τη συμπερίληψη των ανθρώπων με αναπηρία και δεν μπορώ να μην αναφέρω μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την 20η επέτειο του Φόρουμ φέτος να σας συγχαρώ και για την δουλειά που έχετε κάνει για να προβάλλετε τα θέματα αναπηρίας. Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω και άλλα μέλη της κοινωνική πλατφόρμας που εργάζονται στο θέμα της αναπηρίας σε παροχή υπηρεσιών Inclusion Europe, αυτισμό στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την ε, Επανένταξη και άλλα μέλη τα οποία εργάζονται για την συμπεριλήψη των ατόμων με αναπηρία. Η κοινωνική πλατφόρμα υφίσταται για να δώσει δύναμη, κάνοντας τη σύνταση μεταξύ του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη όλων των ομάδων που αντιμετωπίζουν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ανισότητα στην κοινωνία μας. Και βλέπουμε ότι αυτές οι ομάδες υποεκπροσωπούνται έντονα σε τόπους και μέρη και όπου υπάρχει ιδρύτερη εξουσία και χρήματα. Ένα από αυτά τα μέρη είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που σας συνεχάρισαν για τη δύναμή σας να βρίσκεστε εδώ σήμερα σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οίκο Ευρωπαϊκής Εξουσίας. Θέλουμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή κοινωνία όπου όλοι θα αναγνωρίζονται για την ξεχωριστή τους συνεισφορά ανεξάρτητα από την ηλικία την εθνικότητά, το φύλλο, την ηλικία, την αναπηρία τους. Εγώ προέρχομαι από μια ένωση για τα δικαιώματα των παιδιών. Έχω εργαστεί 12 χρόνια για, στο Eurochild, ένα δίκτυο το οποίο προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών. Για μένα λοιπόν το να δώσουμε στα παιδιά από νεαρή ηλικία την δυνατότητα να έχουν σαφή αντίληψη της ταυτότητάς τους στη ζωή είναι κλειδί. Και πιστεύω ότι αν από την παιδική ηλικία εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στον καθένα για αυτό που πραγματικά είναι, ανεξάρτητα από τις ικανότητές μας, θα σχηματίσουμε ενήλικες οι οποίοι σε, κατά πάσα πιθανότητα θα φοβούνται λιγότερο τους άλλους και θα είναι πιο ανοιχτοί στο οποιοδήποτε διαφορετικό στοιχείο. Το σλόγγαν ε, «Τίποτα για μας χωρίς εμάς» είναι πολύ δυνατό και προϋποθέτει ότι τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ισχύω, όπου και αν βρίσκονται, είτε στην οικογένεια, είτε η παροχή υπηρεσιών, είτε στην πολιτική ζωή, να ζητήσουμε από εσάς και να ευχαριστήσω τους βρεβουλευτές ε, εδώ, γιατί κυρίως την κυρία Χάρκιν, να πείτε κι εσείς για λίγο στη θέση των ανθρώπων αυτών που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Σημαίνει ότι τα άτομα σε θέσεις εξουσίας θα αφιερώσουν χρόνο για να κατανοήσουν και τις θέσεις και τις ανάγκες των όσων υποστηρίζουν. Και τέλος, ο ρόλος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα αυτά τα οποία υποστηρίζουμε θα πάνε σε ένα μέρος, σε μια κατάσταση που θα έχουν έλεγχο στη ζωή τους και θα ασκούν τα δικαιώματά τους και την, την, θα καθορίζουν αυτά τη ζωή τους. Μιλάμε για καταμερισμό της εξουσίας, αν θέλετε. Υπάρχουν και άτομα στην Ευρώπη που πιστεύουν ότι είναι μηδενικό το άθροισμα τη εξουσία, ότι αν δώσει κανείς εξουσία θα τη χάσει. Εγώ πάντα θεωρώ ότι η εξουσία είναι σαν την αγάπη. Όσο πιο πολύ έχει κανεί, τόσο πιο πολύ αναπτύσσεται και όσο πιο πολύ δίνει κανεί, τόσο πιο πολύ πάλι αθρίζεται. Πιστεύω ότι το κοινωνικό κίνημα λοιπόν σήμερα στην Ευρώπη βρίσκεται σε μια εξαιρετική στιγμή, σε μια εξαιρετική χρονική συγκυρία. Πριν από κάποιε εβδομάδε η κοινωνική πλατφόρμα κλήθηκε να εκπροσωπήσει την κοινωνία των πολιτών στο Κέτεμπορκ στην ε, σχετική εκδήλωση, όπου συμμετείχαν και πολλά κράτη-μέλη άλλωστε. Και ε, ο κ. Πακλάρκα από το EDF ήταν εκεί και είδαμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να διακηρύσουν τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η πρόκληση δική μας είναι τώρα αυτό να μετατραπεί σε αλλαγή πολιτικής και σε δημόσια επένδυση. Συνολικά, λοιπόν, οι, οι κυβερνήσεις ε, εξέτασαν την ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και για πρώτη φορά, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πραγματικά ένα καθολικό πακέτο συνολικών στόχων που καλύπτουν και την κοινωνική ε, πρόοδο και την περιβαλλοντική πρόοδο και μια βιώσιμη συμμετοχική δημοκρατία. Και όσο προχωράμε προς το τέλος της τρέχουσα στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά έχει την δυνατότητα να εντάξει τους βιώσιμους στόχους στο όραμα της για το μέλλον και στη στρατηγική της για το μέλλον. Φυσικά θα ήταν αφελές να σας παρουσιάσω την κατάσταση ρόδινη. Χρόνια λιτότητας ε, έχουν ε, αποδεκατήσει τα εθνικά κοινωνικά συστήματα και βλέπουμε και φύλακες ε, φτώχειας, αλωτρίωσης, ε, φόβο πολιτικής πόλωσης. Ε, αυτή την περίοδο όμως της αβεβαιότητας και της αστάθειας έχουμε ένα περιβάλλον γόνιμο για αλλαγή, για νέους τρόπους ε, να συνεργαστούμε και να σκεφτούμε από κοινού. Και έχουμε και όλο και πιο πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε αναπτυσσόμενο σώμα, αν θέλετε, νόμων ανθρώπινων δικαιωμάτων τα οποία μπορούμε να προβάλλουμε προς τις κυβερνήσεις μας και να τις ε, καλέσουμε σε λογοδοσία. Έχουμε νέους τρόπους επικοινωνίας που μας βοηθούν να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες, να διαβιβάσουμε καλύτερα το μήνυμά μας. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια αναπτυσσόμενη κοινότητα ανεξάρτητων ατόμων που λαμβάνουν αυτόνομα αποφάσεις, τη φωνή των οποίων δεν θα ε, καταπατηθεί και θα σχηματίσει μια πραγματικά συμμετοχική κοινωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χένσουερθ. Πολύ ωραία η ομιλία σας. Σήμερα στο διάδρομο συνάντησα κάποιον από την Ομίγυρη που μου είπε θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον, να μην παρελθοντολογούμε, να μην ε, ε, αναμασούμε το παρελθόν και πώς ζούσαμε πριν από 20-30 χρόνια. Να κοιτάμε το μέλλον. Αναφερθήκατε στα παιδιά και είπατε πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργήσουμε στα παιδιά ε, αυτοπεποίθηση και όταν συναντούν κάποιον με αναπηρία να μην εκπλήσονται είναι να μην τους ξενίζει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαπαιδαγώγηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μάουρο Δωτής, μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών. Honorable Stevens, signora Anka. Κυρία Stevens, κυρία Άνκα, Επίτροπε Άισεν, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ πρόεδρε Βαρδακαστάνιο, και εγώ Έχω ξαναεπισκεφθεί αυτό το ημικυκλό. Ποτέ δεν το έχω δει τόσο γεμάτο, δεν έχω δει ποτέ και τόσο όμω χαμόγελο όπω αντικρίζω σήμερα. Και για αυτό το λόγο σα ευχαριστώ που καλέσατε την Επιτροπή των Περιφερειών και εμένα εν ονόματι του πρώτου κυρίου Λάμπερτ. όπως ξέρετε, οι κοινότητε και οι περιφέρειες έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτική απασχόληση, κατάρτιση γενικότερα στα κοινωνικά. Και ε, πρόσφατα θα έχουμε συζητήσει αυτά τα του κοινωνικού πυλώνα. Εγκρίθηκε αυτός και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για όλους να υπάρξουν εγγυήσεις εξισορρόπησης της ιδιωτικής με την ε, ε, επαγγελματική ζωή. Κανείς να μην μείνει πίσω. Είναι βασικός στόχος μας. Επίσης έχουμε συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε για τους ανθρώπους με αναπηρία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν εμπλακούν περιφερειακές τοπικές αρχές και θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση οι Ευρωπαίοι. Επομένως, χρειάζεται καταλήγουμε να προγραμματίσουμε τους ε, πόρους που θα πρέπει να επαρκούν. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν χρηματικοί πόροι αλλά και μία υπευθυνότητα και έτσι να υπάρχει ποιοτική αρρωγή. Πρόκειται επίσης και για το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη και μειώνεται το εργατικό δυναμικό και αυξάνουν οι πιο ηλικιωμένοι. Μέσα σε λίγα χρόνια πρόκειται να δούμε μεγαλύτερη αύξηση, μεγαλύτερη γύρανση του πληθυσμού. Θα σας τα λέω, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτική συνοχής είναι ζωτική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό, για τις ε, πόλεις μας, της περιφέρειές μας, για όλη την Ευρώπη. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά τις ε, επενδύσεις που ωφελούν τους ε, Ευρωπαίους όταν αξιοποιούνται. Και το πιο σημαντικό όσον αφορά τα μέσα χρηματοδότησης είναι το να φροντίζουμε την απασχόληση και να χρησιμοποιούμε το κοινωνικό ταμείο στη χώρα μου το κοινωνικό ταμείο επιτυχώς έχει χρηματοδοτήσει κάποιες πρωτοβουλίες και νομοθετικά έχει κατοχυρωθεί το ότι δεν είναι δυνατόν να μην είναι προτεραιότητα η πλαισίωση των ανθρώπων με αναπηρία. Οπότε και έχουμε ολόκληρες οικογένειες που έχουν το πρόβλημα της αναπηρίας και βοηθούνται τα παιδιά του να πάνε στο σχολείο, γιατί όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα δεν μπορούν να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Άρα θα πρέπει να συνεχίζεται η χρηματοδότηση, επομένω. Απερίφατα θα σα λέω ότι είχε 100% δίκιο η Επίτροπο όταν λέει ότι θα πρέπει να προβούμε σε κάποια αποφασιστική πολιτική επιλογή. Και ελπίζω ότι αυτά τα οποία είπε η Επίτροπο θα τα αγκαλιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να υπάρχουν επομένω επαρκή σπόρ για την κοινωνική πολιτική. Περί αυτού πρόκειται και χωρί να έχουμε την εκταμείευση ικανών πόρων, τότε πώς θα κατοχυρωθούν τα σχετικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Θα μείνουν λόγια κενά όλα αυτά τα οποία εξαγγέλουμε και θα πρέπει να υπάρξει όσο γίνεται περισσότερη ευελιξία για να βοηθήσει η Ευρώπη όποιον έχει ανάγκη. Όχι μόνο στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού και θα πρέπει να δούμε τι μορφή θα πάρει αυτή σας η απόφαση, αυτή σας πρωτοβουλία κύριε Επίτροπε όσον αφορά το Ταμείο Ανθρώπινου Δυναμικού. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι έχει αγκαλιάσει πραγματικά ε, τον κοινωνικό πυλώνα η Επιτροπή μας. Και έχουμε κάποιες συμπολίτες μας που έχουν ε, στείλει ένα γράμμα και είπε αγαπητοί ε, οι υπουργοί έχουμε πρόβλημα επιβίωσης, έχουμε αναπηρία και έχουμε πρόβλημα και συμμετέχουμε στην κοινωνική ζωή μόνο μέσω της προσωπικής βοήθειας. Οπότε μόνο ε, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Περιφερειακή Αρχή είναι να βοηθήσει, όχι να δώσει ελεημοσύνη. Θα πρέπει επομένως να γίνουν σεβαστά αυτά τα δικαιώματα, αυτά τα οποία προτάσσονται σε αυτή την επιστολή. Δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε κατά μέρους αυτούς τους ανθρώπους. Και οπότε βλέπουμε το πρόβλημα δεν είναι ιατρικό, είναι κοινωνικό. Επομένως τέτοια προσέγγιση χρειάζεται. Έτσι θα κάνουμε τις πιο σωστές επιλογές για την περίοδο μετά το 2020. Σας ευχαριστώ, κυρία τη, Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κούνεβα, Ευρωβουλευτή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Χέλγα. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλωσορίσατε στο σπίτι σας. Λέω σπίτι σας, γιατί εδώ είναι το κέντρο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας όπως όλα τα σπίτια, έχει και αυτό τα προβλήματά του. Μην κοροϊδευόμαστε, αλλά έχει γερά τεμέλια της αξιοπρέπειας, της ισότητας, της διαφορετικότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Πολλές φορές κάποια από τα τεμέλια τρίζει και εμφανίζει ραγμές. Στόχος όλων μας θα έπρεπε να είναι η τωράκισή του. Και εσείς πιστεύω πως συμβάλλετε ενεργά. Το αποδεικνύετε σήμερα με την παρουσία σας. Παρά τις δυσκολίες που είμαι σίγουρο ότι συναντήσατε, βρίσκεστε εδώ για να εκπροσωπήσετε την Ευρώπη της διαφορετικότητας. Και εγώ με τη σειρά μου βρέθηκα εδώ για να εκπροσωπήσω εμάς που η φωνή μα πολύ συχνά δεν ακούγεται και δεν φτάνει στα κέντρα λήψη αποφάσεων. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τη ζωή μα. Ρωτάω λοιπόν την Κομισιόν και το Συμβούλιο πόσο νομίζουν ότι αξίζει η ζωή μα, γιατί αν κρίνω από τα κονδύλια που διαθέτουν για εμάς τα άτομα με αναπηρία τη τιμολογούν πολύ φθηνά αν όντω θέλουν μια κοινωνική Ευρώπη, πρέπει να κάνουν τουλάχιστον δύο πράγματα. Πρώτον, να σταματήσουν τις πολιτικές λιτότητας. Δεύτερον, να χρηματοδοτήσουν με ανάλογα κοντήλια τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγική για την Αναπηρία. Αλλιώς οι πολιτικές αυτές είναι ανέξοδες ευχές. Και είναι καιρός να μπει να μπει τέλος σε υποκρισία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα. Όντως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε ένα πολύ αγαπητό συνάδελφο από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, τον κύριο Ροδόλφο Κατάνη. Ευχαριστώ και καλησπέρα. We have a challenge. Υπάρχει μπροστά μας μια πρόκληση. Να σας πω δηλαδή κάτι σημαντικό χωρίς να αναλώσω πολύ από το χρόνο σας. Είμαι τυφλός και έχω ένα ειδικό ρολόι και με την αφή τώρα διαπιστώνω ότι ήδη έχω αναλώσει 20 λεπτά από τον χρόνο που έχετε δώσει στους προσκεκλημένους να μιλήσουν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο άβολα νιώθω πάντως. Θα πρέπει να σας πω ότι το φόρουμ μας έχει ετοιμάσει ένα σημαντικό έγγραφο που αφορά την μέλουσα Ευρωπαϊκή Στατική για τα πρόσωπα με αναπηρία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε μέσα σε 5-6 λεπτά και όχι περισσότερα να σας τα πούμε. Όχι, δεν θα σας πω θεωρητικολογίες κάποια πραγματικά περιστατικά θα σας παρουσιάσω. Τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για μας. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να μάθουμε τι μορφή θα έχει. Και επιθυμούμε έγκληση στους ηγέτες να εγκρίνουν μια στρατηγική η οποία θα καλύπτει τα εξής. Και δεν είναι πολλά αυτά να καλύψει ό,τι προβλέπει η σύμβαση του ΟΗΕ με μια προοικοδότηση που να καλύπτει την υλοποίηση και επομένω να υπάρχει και η δημοσιονομική πρόβλεψη για την εποπτεία της εφαρμογής και όλα αυτά να έχουν σχέση με την υλοποίηση της στρατηγικής του 2020 ούτως ώστε να υπάρχουν κάποια ευφύς αντιμετώπιση και εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα και όλα αυτά στα πλαίσια τη θεματολογία του 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη και τους σχετικούς στόχους και να βασίζεται στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα πρόσωπα με αναπηρία και έτσι να εμπλέκονται όλα τα θεσμικά όργανα, όλες οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την ε, εποπτεία της εφαρμογής, την υλοποίηση τελικά της στρατηγικής, οπότε θα πρέπει αυτή η στρατηγική να είναι η ατμομηχανή για, αυτήν, για αυτό το θεματολόγιο 2020-2030 και όπως ήδη είπε ο Πρόεδρος να καλύπτεται και να προβλέπεται το 2021 ως ε, έτος για τους ανθρώπους με αναπηρία που είναι σημαντικό. Επίσης, απευθυνόμαστε στους Ευρωπαίους ηγέτες ώστε να μπορέσουν να προβλέψουν τις εξής δράσεις στα πλαίσια της στρατηγικής 2020-2030. Α, 16-16 είναι οι προτάσεις μου και τα σημεία που θέλω να ε, σταθώ. Αλλά θα είναι πάρα πολύ σύντομος. Να ε, κυρωθεί το προαιρετικό πρωτόκολλο της ε, σύμβασης του ΟΗΕ. Έχει καθυστερήσει η Ένωση. Θα πρέπει να καλύψει το χαμένο χρόνο. Και θα πρέπει να προβλέπεται ένας διαδρομένος διάλογος με τις ε, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των προσώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους και να προβλέπεται ένα κονδύλι στον προπολογισμό για αυτού του είδους την συμμετοχή, τη διαβούλευση και χωρίς χρήματα τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Ούτε καν λειτουργία δεν μπορεί να κάνει ο παπάς αν δεν έχει τον οβολό μας. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, διοργανικός μηχανισμός ε, συντονισμού και να δούμε πού μπορεί να εστιάσει τις προσπάθειες του κάθε θεσμικό όργανο, κάθε ευρωπαϊκή υπηρεσία, ακριβώς όπως προβλέπεται στο άρθρο 23, παράγραφος 1 της ε, σύμβασης του ΟΗΕ. Θα πρέπει να εποπτεύεται η υλοποίηση των ε, επιπτώσεων για τις πολιτικές, για τα προγράμματα, ούτω ώστε να υπάρχει συμμόρφωση και να είναι σύντονα όλα αυτά με την σύμβαση του ΟΗΕ. Επίσης θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την δήλωση των αρμοδιοτήτων ούτω ώστε να καλυφθούν όλες οι πολιτικές, όλοι οι τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κάποια μέτρα. Θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε αυτόν τον κατάλογο το υπήν των αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει επίσης να δούμε το πώς δεν θα υπάρχει διάκριση εις βάρος των προσώπων με αναπηρία. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες που υπάρχουν, που αναγνωρίζονται για αυτούς δηλαδή που δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στον κοινωνικό βίο. Θέλουμε και αυτόν τα δικαιώματα να αναγνωριστούν και θα πρέπει αυτά όλα να συμμετοχθούν σε κάθε δράση της εν λόγω στρατηγικής. Θα πρέπει να έχουμε νομοθεσία για να μην έχουμε διάκριση δυσμηνή με εφορμή την αναπηρία και αυτό να μην έχει ε, εγκάρσιο χαρακτήρα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κάποιο είδους μηχανισμοί προς τούτο. Επίσης να έχουμε κάποιο είδους ε, εκστρατεία σφαιρική, γενική και να υπάρξει συνειδητοποίηση του, του, του, του, των, των όσων επιτάσσει η σύμβαση του ΟΗΕ να καταπολεμούνται έτσι εσμενείς διακρίσεις για αυτούς που έχουν αναπηρία γιατί δεν μπορείτε φανταστείτε πόση αναπηρία επικρατεί παρά όλα τα ωραία λόγια που τόσο συχνά έχουμε την ευχαρίστηση να ακούμε. Θα πρέπει να και κάποιο είδου κατάρτιση, εκπαίδευση για όλο το προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλου που δουλεύουν εδώ όσον αφορά τη σύμβαση του ΟΗΕ για την ε, προσέγγιση βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσβαση σε υπηρεσίες κλπ. από πλευράς των ε, προσώπων με αναπηρία. Και τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις για κάποιες πολιτικές σε τομείς κατεπήγοντες όπως ας πούμε κάποιους πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν αναπηρία την δικαιοπαιδική του ικανότητα, ε, εμπλοκή στην λήψη αποφάσεων, ε, στην ασφάλειά τους και θα πρέπει έτσι να ενταχθούν, να στην ε, κοινωνία, να αξιοποιηθούν έτσι κάποιοι κοινοτικοί πόροι, τόσο ώστε να βοηθήσουμε να υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες για αυτούς από πλευρά των κοινοτήτων. Σχεδόν τελείωσα. Ε, νομοθεσία επίσης, ούτως ώστε να βοηθήσουμε την προσβασιμότητα και μέσω της πράξης προσβασιμότητας και θα πρέπει επίσης η προσβασιμότητα να είναι προαπαιτούμενο, προϋπόθεση σε κάθε προγράμματα σε κάθε πρόγραμμα συγγνώμη, που τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτεί χωρί κανένα συμβασμό. Και επίση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή τη κείμενη νομοθεσία για την προσβασιμότητα. Όπω α πούμε η προσβασιμότητα σε, κιν, σε κινητές εφαρμογές και το ίντερνετ γενικότερα και να βοηθήσουμε τι πρωτοβουλίε για την ελεύθερη διακίνηση να προσώπων μια τα δικαιώματα των ε, επιβατών επίσης, την φορητότητα των υπηρεσιών και επίσης να έχουμε κάποιο είδους ε, έγκυρα αποτελεσματική κάρτα για το μια αναπηρία. Επίσης θα πρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που προβλέπει η Σύμβαση του Τέλος, να υπάρξουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να είναι εγγυημένο το ότι τα θεσμικά όργανα, οι υπηρεσίες, οι πρωτοβουλίες είναι προσβάσιμες σε πρόσωπο αναπηρία και το ότι αυτή η προσβασιμότητα συστηματικά τηρείται με κάποιο είδους γενική, σφαιρική προσέγγιση. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. είναι δύσκολο και για τα κρατημέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει όλα αυτά και για αυτό και χρειάζεται μια νέα στατική τα πώς είναι απειρία για την περίοδο 2020 έως 30. Δεν μου είναι εύκολο να σας πω τι σκέφτεται το φόρουμ για την ισχύουσα τώρα στρατηγική για τα πρόσφατα με αναπηρία. Γενικώ μιλώντας δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι πολλές από τις προβλεπόμενες δράσεις δεν έγιναν ή δεν επιέζαν τόπο. Και δεν βλέπουμε μέσα στην σημερινή δύσκολη κατάσταση να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτω ώστε στο λίγο χρόνο που απομένει αυτό το οποίο πάσχει να διορθωθεί πάντως. Άκουσα. Δύο τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες της ε, Επιτρόπου Τάιζεν και ελπίζουμε ότι τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει τα υπεσχημένα. Ποντάρουμε στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα, πράγματα είναι πιο δύσκολα με τα κράτη-μέλη, έχουμε λιγότερη εμπιστοσύνη το υπήρνει σε αυτά, αλλά είπαμε υπάρχουν μέλουσε υποσχέσει στο μέλλον, αλλά και επιτυχία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο τμήμα της ε, του πανελ Θα δώσω το λόγο αυτό τώρα στο κοινό. Δυστυχώ δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μα και θα ήθελα λοιπόν να είμαστε όλοι πολύ σύντομοι. Ο επόμενο λοιπόν που θα πάρει το λόγο είναι η κυρία Πιέρο Γκριφό. Πού βρίσκεται όμω. Okay. Good morning. Bonjour. Καλημέρα σα. Και εγώ να σας μιλήσω εκ μέρους του Ιταλικού Φόρουμ. Έχουμε 300.000 και 800 εκατομμύρια από φτωχού, από περιθωριοποιημένους στις αντισόμενες χώρες. Να σας διακόψω. Το 2... Η θέση έδρανα 298 για να μπορέσει να σα βρει η κάμερα. Μιλιώνει τη 700 εκατομμύρια είναι τα πρόσωπα με αναπηρία που πολλέ φορέ βοηθούνται μόνο από δωρεέ, δωρεέ κρατικέ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο μεγάλο δωρητής προ αυτού τους ανθρώπους. Και η Επιτροπή του ΙΕ ε, έχει προσπαθήσει τελευταία ούτω ώστε να προσφέρει σε αυτά τα πρόσωπα μια βοήθεια. Και υπάρχουν αυτέ οι τελικέ συστάσει του άρθρου 11 και του άρθρου 32 τις σύμβαση που αφορούν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια και την σχετική συνεργασία. Και επίση αναφέρεται μια σειρά συστάσεων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και εδώ να επενθυμίσουμε το τι γίνεται, το πόσο σημαντικέ είναι αυτέ οι δράσει για αυτά τα πρόσωπα. Και θα πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο να τηρήσουμε τα όσα προβλέπονται και θα πρέπει όλοι να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Πολλές φορές όμως δεν υπάρχει το σχετικό πλαίσιο. Πολλές φορές δεν βοηθούνται οι οργανώσεις αυτών των προσώπων πολλές φορές δεν υπάρχουν οι πόροι. Ή δεν φτάνουν σε αυτές τις τρίτες χώρες ή δεν διατίθενται για τα πόσο με αναπηρία. Οπότε χρειάζεται μια στρατηγική σε σχέση με, την, με αυτή την ανοιξιακή πολιτική που να καλύψει τα πρόσωπα με αναπηρία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο λακωνικός. Θα ήθελα και από τους υπόλοιπους ομιλητές να θέλω να παρακαλέσω να τηρήσουν το χρόνο αγόρευσης. Ο κύριος Τζον Ντόλ έχει το λόγο από την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία της Ιρλανδίας. It I'm very honored. John Dolan. Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι επικεφαλής μιας ε, πολύ ισχυρής ε, Ιρλανδικής Αντιπροσκοπίας. Περίπου 300.000 ε, άτομα με αναπηρία δολοφονήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς, γιατί οι ναζιστές τους θεωρούσαν ως ανάξιους να ζουν τους ανθρώπους με αναπηρία. Και μάλιστα αυτό το σχέδιο αποδεκατισμού των ατόμων με αναπηρία εύκολα εφαρμόστηκε το 1948, μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη ε, με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκε το δικαίωμα που έχουν οι άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή είναι ανθρώπινα πλάσματα, χωρίς τίποτα παραπάνω. Και μάλιστα έξι δεκαετίες μετά τα Ηνωμένα Έθνη θέσπισαν τη σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η σύμβαση αυτή είναι μια αναγνώριση ότι τα Ηνωμένα Έθνη και οι χώρε που υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή, συμπεριλαμβανομένη τη Ιρλανδία, δεν είχαν ε, βελτιώσει επαρκώς ε, τη ζωή, την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στην επικράτειά τους δεν είχαν γίνει ακόμη κάτοχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτά τα άτομα, δεν είχαν ακόμη κατοχυρώσει την αναξιοπρέπειά τους, δεν είχαν εθαρρυνθεί να εκπληρώσουν το δυναμικό τους και να συμμετέχουν. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι τμήμα του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία είναι σημαντικό και ζωτική σημασία σε εργαλείο για να υλοποιήσουμε αυτή τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία. Βέβαια, η εκφώνηση διακηρύξεων δεν σημαίνει έμπρακτη εφαρμογή. Όταν ήμουν ε, νέος, ε, ζήγησα πολλά, πολλά γουρούνια. Αλλά βέβαια το να ζυγίζει κανείς ένα γουρούνι δεν σημαίνει ότι αυξάνει το βάρος του. Χρειάζονται έργα και όχι απλώς λόγια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας δημοκρατικός φορέας, ένα δημοκρατικό θεσμικό όργανο σε πολυτάραχους καιρούς και ταραγμένο κόσμο. Αυτό είναι αναφυσβήτητο. Και αν δεν ασκήσετε εσείς την ηγετική, μας, την ηγετική σας ικανότητα, θα μας αφήσετε εσκεμένα στο περιθώριο, να μαραζώνουμε. Εν κατακλείδη θα ήθελα να απογνωρίζουμε την τελευταία δεκαετία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει με πυγμή, με αποφασιστικότητα, με κύρος και με αποτελέσματα. Θέλουμε εδώ και τώρα να δούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα αυτή την πυγμή, αυτή την αποφασιστικότητα που θα τη μεταφέρουν στην καθημερινότητα αυτών των 80 εκατομμυρίων συμπολιτών μας με αναπηρία και των οικογενειών τους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος μας ομιλητής είναι ο Σλάβο Μιρ Μπεσόφσκι. Παρακαλώ να είστε σύντομος ώστε να προλάβουν όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο να μιλήσουν. Ο κύριος Σαβόμιρ Μπεσόφσκι από το Κέντρο Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία. Σας ευχαριστώ θερμά, λέει ο κύριος Μπεσόφσκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους διοργανωτές για την εκδήλωση αυτή και να αφιερώσω την στοργή μου σε εκείνους τους ε, συμπολίτες μας που δεν μπόρεσαν να έρθουν, που έμειναν ε, κλεισμένοι σε τέσσερις στίχους, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα ε, και το πάνελ, κυρίως ε, τον πρόεδρο του ETF και τους συντονιστές αυτής της συζήτηση. και να ευχαριστήσω θερμότατα και την κυρία Χάρκιν που έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή και για τη δική μου ομιλία, όπως και ο κύριος Μάουρο Ντατής. Η κυρία Χάρκιν είπε ότι προσέλαβε ένα άτομο με αναπηρία πρόσφατα και μόνο τότε συνειδητοποίησε τι σημαίνει η καθημερινότητα του ατόμου με αναπηρία. Ε, και ε, Μάλιστα, πολλές φορές ε, ένας άνθρωπος με αναπηρία δεν ελπίζει καν να βρει θέση εργασίας, γιατί πολλοί θεωρούν ότι η Βρυξέλλες είναι ένα απρόσιτο μέρος και Μπορεί να πιστεύει κάποιο Πολωνό, α πούμε, με αναπηρία, ότι καλύτερα η Βαρσοβία είναι πιο κοντά από ότι οι Βρυξέλλε που τη νιώθει ω κάτι πολύ απόμακρο. Μα ρωτήσατε εμπράκτο ε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, γιατί έχουμε την νομοθετική πράξη για την προσβασιμότητα. Αλλά στο άρθρο 19 ε, της ε, σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τα γενικά σχόλια που είχαμε πρόσφατα για το άρθρο 19, διαπιστώνουμε ότι ε, το πεδίο εφαρμογής ε, του άρθρου 19 είναι πολύ ευρύτερο. Ε, και επίσης μιλούμε για την προσωπική αρρωγή, γιατί χωρίς προσωπική συνδρομή ούτε οι συνάδελφοί μου, ούτε όσοι βρίσκονται υπό την κυδαιμονία ή την επιτροπή των συγγενών ή κάποιων άλλων ε, ή κάποιοι που θέλουν να βρουν μια δουλειά δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Γιατί η ζωή είναι θεμελιώδες και αναπαλωτρίο το δικαίωμα και θα πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι. Η στρατηγική λοιπόν χρήζει πιο τακτικής, πιο συχνής αξιολόγησης με συγκεκριμένους και προσδιορισμένους δείκτες που δεν θα ε, λαμβάνει μόνο υπόψη το βιωτικό επίπεδο ή τη υγειονομική περίθαλψη, αλλά και την απαραίτητη κοινωνική υποστήριξη και υποστήριξη που πραγματικά θα εξασφαλίζει την άσκηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων για να είναι πραγματικά ανεξάρτητα και αυτόνομα στη ζωή τους. Μην βιάζετε να χειροκροτήσετε. Θα ήθελα να σας αναφέρω ε, και μία φράση από την από μια ε, πρόεδρο ε, της αντιπροσωπείας της ε, Ένωσης Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση. Αυτή την ερώτηση δεν θέλω να σας μεταφέρω. Είστε έτοιμοι για τη σύμβαση. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω μεταφέροντας τα λεγόμενα της Προέδρου. Ευχαριστώ. Κον. Ο Βασίλειος Κουτσιάνος έχει παρακαλώ τώρα το λόγο από την Ελλάδα. Παρακαλώ να είστε σύντομος κι εσείς. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλης Κούτσιανος και είμαι υπεύθυνο διεθνών σχέσεων της Ελληνικής Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο φορά εκπροσώπησης των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρου Ατόμων με Αναπηρία. Βρίσκομαι εδώ γιατί θέλω να εκφράσω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του συνόλου των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία και των οικογενειών τους που τα τελευταία οχτώ χρόνια αγωνίζονται αδιάκοπα προκειμένου να ανατρέψουν τις διμενείς καταστάσεις που βιώνουν από τα συνεχιζόμενα μέτρα λιτότητας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά και με όλη τη δύναμή μας για την άρση των μνημονιακών μέτρων που έχουν επιφέρει μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις μας, καθώς και για την αποτροπή εφαρμογής οποιοδήποτε μέτρο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση των αναπηρικών επιδομάτων και στη μείωση της χρηματοδότησης δομών και προγραμμάτων που προωθούν την κοινωνική ένταξή μας. Αγωνιζόμαστε ενάντια στη φτωχοποίηση, στην εξαθλίωση και σε οποιοδήποτε περιορισμό των ανθρώπινων και συνταγματικά ακατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των απαιτήσεων της Σύμβασης του Οργανισμού Ενωμένων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω είναι πως σε όλη αυτή τη τιτάνια προσπάθειά μας τα θεσμικά όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να είναι δίπλα στο ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα και τις διεκδικήσεις του διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε όλοι μαζί από κοινού να διασώσουμε τις αξίες που στηρίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό αρχές όπως είναι η αξιοπρέπεια ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ισότητας της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. ως εθνικό αναπηρικό κίνημα ζητούμε με όλη τη δύναμή μας από την ευρωπαϊκή ένωση να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία που θα προωθεί την εφαρμογή της σύμβασης των ηνωμένων εθνών και θα βελτιώνει στην πράξη την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγαλύτερη θεσμική και πολιτική ευάνθυνση που σχεδιάζεται στις μέρες μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εργαστούν σκληρά σε συνεργασία με το Εθνικό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία για την εφαρμογή μιας κοινή ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής που θα αντιμετωπίζεται με αναπτυξιακή διάσταση και όχι ως οικονομικό βάρος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στον κύριο Μάρκου Γιώκινεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοφών. Συγγνώμη, κυρία. Μάλλον κύριο, Εκπροσωπώ τον, την Ευρωπαϊκή Ένωση Κοφών. Είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοφών και εκπροσωπώ και τους χρήστες της νοηματικής στην Ευρώπη. Θα σας παρουσιάσω την προπτική των κοφών, τη σκοπιά των κοφών για την Ευρω... μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναμυρίες. αναπηρίες. Τα καταληκτικά συμπεράσματα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ε, στάθηκε σε δύο ζητήματα και αυτά εντόπισε. Το ένα αφορά την ελευθερία έκφρασης και γνώμης και την πρόσβαση σε πληροφορίες και το δεύτερο είναι η συμμετοχή στον ε, πολιτικό και δημόσιο βίο. Η Επιτροπή λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών σύστησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να επιβάλλει την εφαρμογή της νομοθεσίας που επιτρέπουν την πρόσβαση στην ενημέρωση και την πληροφορία. Με την Ευρωπαϊκή Νομοθετική Πράξη για την Προσβασιμότητα έχει προταθεί ότι δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή την νομοθετική πράξη να καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες ώστε να σημειώσουμε έτσι πρόοδο και να βελτιώσουμε πραγματικά την προσβασιμότητα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Πολύ συχνά η κοινότητα των κοφών ε, και των χρηστών της νοηματικής μένουν στο περιθώριο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες ε, με βάση τα συμπεράσματα της Ειδικής Επιτροπής ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ και να εξασφαλίσουμε και μία παρακολούθηση του ρυθμού εφαρμογής αυτής της στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η συμμετοχή στον πολιτικό και δημόσιο βίο των ατόμων με αναπηρία. Μην ξεχνάτε ότι η προεκλογική περίοδος έχει κύρια σημασία γιατί δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες και επιτρέπει στον κόσμο να ψηφίσει έχοντας γνώση της κατάστασης. Οι πληροφορίες αυτές λοιπόν θα πρέπει να είναι προσιτές ε, και στους κοφούς με την νοηματική και όλο το υλικό αλλά και οι πολιτικές αναμετρήσεις ε, να είναι προσιτές και στους κοφούς και χρήστες της νοηματικής. Να προσαρμόζονται λοιπόν όλα αυτά τα υλικά στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των κοφών. Σας ευχαριστώ. Paldies, Zāra. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή. η κυρία Ζάρα από τον εμένα Βασίλειο. Um, I am the director of... Είμαι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την ανεξάρτητη διαβίωση και έχω μία ερώτηση να κάνω. Πώς οι άνθρωποι αμφισβητούν το δικαίωμά τους και τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες παρά την ε, η ύπαρξη της ε, συνθήκης του ΟΗΕ, το τελευταίο έτος φαντάζομαι ότι κάθε άτομο με αναπηρία που κάθεται εδώ στην αίθουσα αυτή έχει νιώσει να αμφισβητούνται τα δικαιώματά του. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη που χρειάζονται προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα όσα μπορεί να τους προσφέρει η χώρα τους και η Ευρώπη. Τμήμα αυτών είναι η πρόσβαση σε μέτρα όπως ε, για παράδειγμα η νοηματική, η διερμηνία και ο, η προσωπική βοηθή να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό κάθε ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και όχι μόνο σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται συγκεκριμένα της αναπηρίας. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά διαρθωτικά ταμεία θα χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλίσουν την συμπερίληψη όλων των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να δρουν ως άτομα και πλήρεις πολίτες στην κοινωνία τους, στην κοινότητά τους, προκειμένου να έχουμε πλήρη έλεγχο στη ζωή μας. Τα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υποστορχθεί καθολικός σχεδιασμός σε βασικές υποδομές προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη πιο προσβάσιμη σε όλους. Θέλουμε η συμπερίληψη στις κοινότητές μας να είναι αυτόματη, όχι προϊόν αγώνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Γκραπίνη, Ευρωβουλευτής. Η κυρία Γκραπίνη. Εδώ βρίσκομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει η κυρία Γκραπίνη. Πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένη. Είμαι εντυπωσιασμένη από αυτά που βλέπω και διαπιστώνω ότι συμβαίνουν εδώ σήμερα. Συγχαίρω τους ε, διοργανωτές και σας συγχαίρω και εσάς προσωπικά, γιατί εσείς γνωρίζετε τα δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να έχετε. Είσαστε δεκάδες εκατομμύρια. Ακολουθήσα την πρόσκληση λοιπόν αυτή που έλαβα από την διακομματική ομάδα για τα άτομα με αναπηρία γιατί στη χώρα μου έχω ασχοληθεί πολύ με ενώσεις ε, ατόμων με αναπηρία, άτομα τα οποία ήταν άριστα ενταγμένα στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για άτομα τα οποία δεν μπορούμε να μην τα αξιοποιήσουμε. Αυτό το ακούσαμε και στην τελευταία παρέμβαση και πιστεύω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματα, τα αυτονόητα τα αυτονόητα. Αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι συνάδελφοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι όσο πιο σωστή, αντικειμενική και διαφανής γίνεται και τα κράτη-μέλη θα πρέπει λοιπόν επιπλέον να κληθούν να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση λοιπόν στα πάντα, στο διαδίκτυο, στην κυκλοφορία, στα κτίρια. Και πραγματικά θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, γιατί και φέτος και φέτος λοιπόν έλαβα θετικέ ε, ειδήσει. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους 751 βουλευτές ε, από οποιοδήποτε πολιτική ομάδα που δεν σας υποστηρίζει και εσάς και τα αιτήματά σας. Σας εύχομαι λοιπόν καλή υγεία, σας εύχομαι ότι καλύτερο και ε, έχετε δικαίωμα σε μια ζωή ακριβώς ίδια όπως ε, όλων των υπόλοιπων. Να μπορείτε να διαβάζετε, να βλέπετε ταινίε, να είστε ενσωματωμένοι στην κοινότητα, να εργάζεστε ανάλογα με τα προσόντα σα και την εκπαιδευσή σα. Σα εύχομαι λοιπόν υγεία πάνω απ' όλα και να είμαστε ενωμένοι εμεί ε, εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω ευρωβουλευτέ να, να ασκήσουμε πίεση στα κρατη προκειμένου εκεί να επιληθούν τα προβλήματα, εκεί που τα αντιμετωπίζετε εσεί, δηλαδή στις πατρίδες σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και κάθε Ό,τι καλύτερο για τις ε, γιορτές. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην ε, Ευρωβουλευτή Ρόζα Εσταράς Φεραγκούτ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι νιώθω μεγάλη τιμή που συμμετέχω σε αυτή την διάσκεψη, σε αυτή την κοινοβουλευτική διάσκεψη με τόσο επιφανεί συμμετέχοντες. Και εγώ είμαι μέλος της διακομματικής ομάδας για, τη, για τα άτομα με αναπηρία. Είμαι αντιπρόεδρος αυτής της διακομματικής ομάδας και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με τα αναπηρία, τους Ισπανούς συναδέλφους από τη ΣΕΡΜΗ και την Όθε, την Εθνική Οργάνωση Τυφλών, που με το έργο τους, με τις προσπάθειές τους μας δίνουν λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση και μας βοηθούν να εμπεδώνουμε όλο και περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έχουμε μια πιο δίκαιη και πολιτική στην Ευρώπη. Επίσης, ήθελα να χαιρετήσω τη σύμμαχό μας στα θέματα της αναπηρίας, την Επίτροπο Τάισεν, που πρωτοστάτησε στην ε, νομοθετική πράξη για τα άτομα με αναπηρίες και την προσβασιμότητα. Ελπίζουμε ότι μετά τους τριμερείς διαλόγους και χάρη στην συμμαχία και τη συνεργασία όλων μας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσουμε αυτή την απαραίτητη νομοθετική πράξη για την προσβασιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, για, για την ε, προσβασιμότητα 2010-2020 έχει πολλά κενά και μάλιστα πρόσφατα στη Μήνη Ολομέλεια συζητήσαμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη μελλοντική μας στρατηγική περιλαμβάνοντας θέματα όπως η προσβασιμότητα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής, μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μία απασχόληση με τις απαραίτητες προσαρμογές, την προσβασιμότητα σε όλους στην ψηφιακή εποχή, την τήρηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ και ούτω καθεξής. Στα λόγια όλοι συμφωνούμε, αλλά χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται προϋπολογισμός, κονδύλια, ε, για να προωθήσουμε αυτές τις δράσεις. Έχουμε και άλλο σύμμαχο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την κυρία Εμίλιο Ράιλι. Επίσης, ε, στην Επιτροπή Αναφορών που συμμετέχω, λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες ε, και παράπονα από κάθε γωνιά της Ευρώπης, από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες που καταγγέλουν τα προβλήματα στην προσβασιμότητα και την αδικία σε τελική ανάλυση που υφίστανται. Γιατί μια ίση δίκαιη Ευρώπη θα πρέπει να είναι μια Ευρώπη προσιτή σε όλους. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω κάτι που το λέω συνέχεια, να το πω και σήμερα. Η παρουσία όλων των φορέων, όλων των συλλόγων, ε, των ατόμων με αναπηρία και όλων ε, που θεωρούμε ότι είμαστε οι εκπρόσωποι τους, θέλουμε να γίνουμε η φωνή σας σε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά που μας είπατε σήμερα από την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία, όπως και από την κοινότητα των ανθρωπίνων, των υπερμάχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να συνενώσουμε τα πνεύματα και τις ψυχές μας και να δώσουμε πραγματική προτεραιότητα στα θέματα και στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Ο επόμενος, η κυρία Στέφανη Γούλιο. Σας ευχαριστώ. Το ΕΝΟΥΣΠ είναι... για το δίκτυό μας, που όσον αφορά τους όσους έχουν ψυχοκοινωνικές ε, αναπηρίες, δυσκολίες. Οπότε θέλουμε να υλοποιηθούν οι συστάσεις. Το πρωτόκολλο στην σύμβαση του ΙΕ να εναρμονιστεί η σχετική νομοθεσία και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εμπλοκή κάποιων οργανισμών που εκπροσωπούν όσους έχουν ε, αναπηρία και τις ε, ψυχοκοινωνικές αναπηρίες επίσης και έτσι να έχουμε ένα πλαίσιο ούτω ώστε να υπάρξει περιεχόμενο στο τη διαβούλευση των διαφορετικών φορέων της Ένωσης και να εμπλακούν οι, όσοι έχουν ε, αναπηρία και άρα χρειάζεται όμως για αυτό το σκοπό και οικονομική υποστήριξη. Για να υπάρχει περιεχόμενο σε αυτό θα πρέπει αυτό το πλαίσιο να ε, οδηγήσει σε κάποιο είδους ε, συναντήσεις, ε, να υπάρχουν κάποιο είδους στοχευμένες ομάδες, εκπροσώπηση των προσώπων αυτών και όχι απλώς να έχουμε ερωτηματολόγια. Ήταν ιστορική η συνάντηση του Ιανουίου 2005 στο Ελσίνκι, τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή το πλαίσιο και όλα αυτά είναι θετικές ε, προϋποθέσεις, προϋποβουλίες μάλλον, αλλά δεν έχουν γίνει αρκετά ούτως ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα όσων έχουν αναπηρία ψυχοκοινωνική. Ε, να μην υπάρχει θεσμής διάκριση μέσω νομοθεσίας για την πνευματική διανοητική υγεία. Να μην εγκλείονται αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι στα νοσοκομεία, να μην υφίστανται ιατρικές αγωγές υποχρεωτικές. Θα πρέπει να εντάσσονται στην κοινωνία και θα πρέπει επίσης να υπάρχει διάγνωση της πραγματικής τους ε, ψυχοκοινωνικής αναπηρίας. Να μην καταπατάσετε το δικαίωμα μας στην ισότητα. Έχουμε πολύ σοβαρές παραδιάσεις ευρωπαϊκών δικαιωμάτων όπως τονίστηκε στην Επιτροπή ε, του ΟΗΕ για αυτή τη σύμβαση από τους ειδικού εισηγητές άρα χρειάζεται όλα αυτά να καλυφθούν από την ε, μέλουσα στρατηγική. Εμείς Περιμένουμε τη βοήθειά σας. Πιέτρο Σιρτσιώνα. Πιέτρο Τσιρτσιώνα είναι ο επόμενος ομιλητής. Το πρώτο που θέλω να σας ζητήσω είναι να υπάρξει αναγνώριση όσον αφορά την κατάσταση της αναπηρίας αυτό είναι η αφετηρία η αναγνώριση των δικαιωμάτων μας. Και αυτή η αναγνώριση ή η μη αναγνώριση είναι κάτι το οδυνηρό γιατί αυτό σοβεί σε πολλά κράτη-μέλη. Και παλιά είχαμε αυτού την πιστοποίηση της αναπηρίας και για να οδηγηθούμε σε κάποιο είδου ε, ωφέλη οικονομικά σκέψη υπηρεσίες ε, στην Ιταλία αλλά σε άλλες χώρες ε, υπήρχε το ίδιο πρόβλημα όσον αφορά τον αυτισμό και πρέπει να εμφανιστούμε σε μια επιτροπή για να μας αξιολογήσει. Και αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε ξανά και ξανά όλη μας τη ζωή. Ε, θα πρέπει να, ε, πρέπει να υπάρχει αναγνώριση ευθύ αμέσω από την γέννησή μας. Έχουμε έρευνα, έχουμε διάφορα πειράματα για τα φάρμακα που μας ωφελούν αυτά όσο πάνε και εντείνονται. Ε, διατίθενται πόροι, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα ηθικά προβλήματα σε σχέση με την φαρμακολογική μακρόπνοη επέμβαση. Αυτά ακόμα δεν έχουν τυχή επεξεργασία. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή μόνο των ιδίων σε αυτή την αξιολόγηση και θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και κάποιες καταχρήσεις, υπερβάσεις από τους γιατρούς και όχι μόνο όσον αφορά τα φάρμακα αλλά για την απόσπαση κάποιες συνένεσης που θα έπρεπε να γίνεται ελεύθερα και συνειδητά παρακαλώ σε όλες τις χώρες όσοι πάσχουν από αυτισμό να ερωτούνται για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η ομιλήτρια δεν καταλαβαίνω καλά, Κουέρβο. Ευχαριστώ, είμαι από την Ισπανία. Μένω στην Ισπανία και συμμετέχω στη χάραξη της πολιτικής και ενημερώνομαι τακτικά για το τι συμβαίνει στο, στο χωριό μου. Μάλιστα συμμετέχω και σε ένα πολιτικό κόμμα και ήμουν και στον ψηφοδέλτη του κόμματός μου στις τελευταίες εκλογές. συμμετέχω τακτικά στη συνεδριάση του πολιτικού, πολιτικού μου κόμματος και στη λήψη αποφάσεων και βοηθώ άλλα άτομα με αναπηρία που έχουν στερηθεί μέχρι στιγμή το δικαίωμα της ψήφου, το δικαίωμα του εκλέγην. Εγώ μπορώ να ψηφίσω. Θεωρώ όμως ότι όλοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου είτε έχουν αναπηρία είτε όχι. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλοί συμβολίτες μου με κάποια αναπηρία που δεν δικαιούνται να ψηφίσουν. Γιατί κάποιοι δικαστές ε, τους στήρισαν το δικαίωμα της ψήφου. Τους κήρυξαν ανίκανους δικαιοπρακτικά. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου ανίκανοι. Είναι πάρα πολύ ικανοί. Μάλιστα, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο άρθρο 29 προβλέπει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τους πολιτικούς τους εκπροσώπους ή να εκλέγονται ως πολιτικοί εκπρόσωποι άλλων ατόμων. Γι' αυτό και θα πρέπει να βιαστούμε ώστε να εφαρμοστεί εμπράκτος η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σε όλες τις χώρες. Θα ήθελα εν τέλει να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης και αυτούς που επέτρεψαν την παρουσία μου εδώ, την Ισπανική Επιτροπή Θέρμη, το κόμμα μου, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας, τους τοπικούς φορείς, όλοι αυτοί συνέβαλαν στο να μπορέσω και εγώ να έρθω στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ώστε όλα τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω θερμά. Thank you so much for your presentation and... Uh, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Επόμενος ομιλητής λοιπόν από την Ουγγαρία. Ντέσι. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, το Ουγγρικό Εθνικό Συμβούλιο για τι Οργανώσει των Ατόμων με Αναπηρία πιστεύετε ότι τα διαφορετικά ταμεία παίζουν ε, ρόλο κλειδί για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι ότι χρηματοποτούν μόνο παρεμβάσεις 30 ε, κοντοετή. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το μετρό τη Βουδαπέστη, παρά το γεγονό ότι ανακαινίστηκε όλη η γραμμή και όλοι οι σταθμοί του μετρό, 8 σταθμοί παραμένουν απρόσβατη για άτομα με, ειδικές, με αναπηρίες. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει ένας υποχρεωτικός μηχανισμός όπου οι ενώσει που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία θα περνάνε πάντα από διαβούλευση προτού γίνονται τέτοια έργα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τέτοιε δραστηριότητε εποπτεία και παρακολούθηση. Στην Ουγγαρία λοιπόν ξεκίνησε μια καινούργια διαδικασία σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία και πώς μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα και όχι σε ιδρύματα, γιατί συχνά οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν, τοποθετούνται σε ιδρύματα, σε χωριά. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να υποστηριχθούν από τα διευθυντικά ταμεία και στο μέλλον και θα πρέπει να υποστηριχθούν και οι προθέσεις τους να ζουν ανεξάρτητα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν άτομα τα οποία ε, χρειάζονται ειδική βοήθεια, ιδιαίτερη βοήθεια και θέλουν να ζήσουν ανεξάρτητα. Πρέπει να διαδοθούν οι καλές πρακτικές και επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά που πάσχουν και υποφέρουν από διάφορες αναπηρίες. Το μηνιαίο τους επίδομα είναι κάτω από 200 ευρώ. Η κοινωνία μας δεν είναι ακόμα απόλυτα συμπεριληπτική. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, πάντα κοιτούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν ο προπολογισμό να συμπεριλαμβάνει πάντα τη διάσταση της αναπηρίας. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής ε, από τη Γαλλία. Mathieu Châtelain. Hi. Uh, dear cousins, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά ξαδέρφια θα έλεγα, γιατί όλοι στην Ευρώπη είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια που έχουμε λάβει χάρη στο έργο των προηγούμενων γενιών είναι το καλύτερο δώρο που έχουμε λάβει ποτέ. Και ένα από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα που έχουμε είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση. Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι θα πρέπει ισότιμα να απολαμβάνουμε αυτό το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης παρά την αναπηρία μας μή θα ήταν δύσκολο για μας να νιώθουμε ότι είμαστε ε, ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα, θα θεωρούμε ότι είμαστε μόνο στα χαρτιά ισότιμοι πολίτες. Στη Γαλλία αναφέρθηκε στην προηγούμενη συζήτηση ότι ότι μπορούσαμε και πριν να γίνουμε Ευρωπαίοι πολίτες να έχουμε τέτοια ελευθερία διακίνηση. Ε, πριν από λίγο ακούσαμε την ομιλία της Επιτρόπου Τάισεν και είχαμε και μια σύντομη συζήτηση μαζί της και πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό το ότι θα επισημάνει αύριο στους ε, υπουργούς την ανάγκη να υιοθετήσουν τη γενική προσέγγιση ώστε να υλοποιηθεί πραγματικά η ελεύθερη διακίνηση και να ληφθεί υπόψη και το θέμα αυτό και στα στις υπηρεσίες υγείας. Και το, το τελευταίο εμπόδιο που συνήθως αντιμετωπίζουμε στις ευρωπαϊκές πολιτικές είναι το θέμα της εφαρμογής. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δείξουν την πραγματική τους βούληση να βοηθήσουν τους πολίτες τους να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους σε πανευρωπαϊκή βάση και ισότιμα. Γιατί Είμαστε πολλές διαφορετικές εθνικότητες στον κόσμο, αλλά έχουμε μία ενιαία ηθαγένεια, την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Σας ευχαριστώ. Thank you so much. The next... Ευχαριστώ. επόμενο ομιλητή από τη Μάλτα. Μάσιμο Ελόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσοι με γνωρίζουν θα γνωρίζουν ότι είμαι αρκετά διστακτικός και σκεπτικιστικός σε ό,τι αφορά τους τόνους χαρτιού που παράγονται από θεσμικά όργανα όπως αυτό εδώ. Και παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος για το κίνημα των ατόμων με αναπηρία και σε ό,τι αφορά τους ηγέτες και σε ό,τι αφορά την διάδραση με τα ίδια τα θεσμικά όργανα, σήμερα το πρωί μόλις Σήμερα το πρωί άκουσα αρκετούς ομιλητές ε, εδώ στην αίθουσα να βασίζουν ε, την ε, ομιλία τους σε μία διάκριση. Εσείς και εμείς και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο λεπτά μόλις, 12 φορές στην ομιλία της είπε εσείς και εμείς. Οι, τα θεσμικά μας όργανα λοιπόν στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πάσχουν. Πάσχουν γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το χάσμα, αυτό το εμπόδιο στην κατανόηση του ότι η ποικιλομορφία δεν σημαίνει εσείς και εμείς. Φανταστείτε να τα λέγαμε έτσι σε ό,τι αφορά τη διατρασή μεταξύ των δύο φίλων, γυναίκες και άντρες, εσείς και εμείς, 12 φορές, σε δύο λεπτά. Να τα λέγαμε αυτά σε σε έγχρωμους, ε, εσείς και εμείς. Αυτό που θέλω να πω τελικά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι το εξή. Πριν από κάποιε δεκαετίε, όταν η ισότητα των φίλων αποτελούσε όνειρο απατηλό, η κοινωνία δημιούργησε πρωτοβουλίε διαφετική διάκριση που έδωσε μια μεγάλη όθηση στις γυναίκες σε μια ανδρακρατούμενη κοινωνία. Δεν έχει έρθει μήπως το πλήρωμα του χρόνου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να κάτσουν να σκεφτούν πώς μπορούν να διαδώσουν ιδέες για μια θετική πολιτική, μια πολιτική θετικών διακρίσεων υπέρ των ατόμων με αναπηρία. Δεν θέλω μόνο στην ομιλία μου σήμερα να σκήσω κριτική κατά των θεσμικών οργάνων και κατά άμα, της Ευρώπης. 70 εκατομμύρια είναι τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν τροπή και άνεδος που εμείς ως κοινότητα των ατόμων με αναπηρία δεν εκλέγουμε πιο πολλούς ε, στο, στις θέσεις αυτές. Έχουμε λοιπόν αριθμητική ισχύ, αλλά δεν έχουμε τους εκπροσώπους μας. Δεν είναι το ξέρετε αυτό. Και ο φίλος μας από την Ευρώπη ανέφερε την αζιστική Ευρώπη. Να θυμάστε ότι αυτή η πόλη στην οποία βρισκόμαστε εδώ αυτό απελευθερώθηκε από το ναζιστικό καθεστώς, από ένα στρατό του οποίου ο επικεφαλής ήταν και ο ίδιος άτομο με αναπηρία. Thank you so much. And next speaker will come. Σας ευχαριστώ. Επόμενος μελητής από τη Γερμανία, ο Γιώαχιμ Ζόιλινγκ. Σας ευχαριστώ. Γιώχη Μιζόλιν ονομάζομαι και μιλώ εξ ονόματος ε, της Γερμανικής Ένωσης Βαρικών. Αυτό που φοβάμαι εγώ, αυτό που φοβάμαι λοιπόν είναι ότι τα άτομα, τα βαρύκοα θα τα ξεχάσουμε στην κατάρτιση των στρατηγικών και στα μέτρα. Και γιατί, γιατί κοιτάξτε για παράδειγμα τους υποτίτλους τους οποίους ε, έχουμε μαζί μας σήμερα. Οι πρώτες ώρες δεν λειτουργούσαν σχεδόν καθόλου και αν ε, κάποιος από εσά προσπάθησε να παρακολουθήσει την όλη συζήτηση μέσω των υποτίτλων, νομίζω ότι δεν θα είχε καταλάβει και πάρα πολλά. Και δεν υπάρχει επίσης και η τεχνή ε, υπότιτλη. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι τεχνικές μας δυνατότητες στην εποχή του ίντερνετ μας επιτρέπουν μόνο να δείχνουμε στα αγγλικά τους υπότιτλους. Δεν είναι αυτό συμπεριλήψη. Και κοιτώντα ε, και το διάλειμμα που κάναμε Πού κάναμε δικτύωση, υποτίθεται ότι θα μιλούσαμε όλοι μαζί από ακουστική άποψη. Αυτό ήταν καταστραφικό και γιατί, γιατί, ξέρετε, 52 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ακουστικά προβλήματα. Σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, φανταστείτε πώς είναι πραγματικά. Και αυτό προφανώς προκαλεί κοινωνικό αποκλεισμό αμα, κατάθλιψη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί τείνουν να απομονώνονται. Γι' αυτό λοιπόν ε, τα προβλήματα ακοής μπορεί να συνεπάγονται μεγάλο πρόβλημα για την υγεία των πολιτών της Ευρώπης και ασκούν μεγάλη πίεση και στο υγειονομικό και κοινωνικό σύστημα άλλωστε, σε περίπτωση που παραμένουν ε, ανεπίλητα. Η σύγχρονη ιατρική παρέχει πολλές δυνατότητες και δεν είναι και δύσκολο να βελτιωθεί η ακουστική μιας αίθουσας. Γι' αυτό λοιπόν οι πολιτικοί ευθύνοντες θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει καλύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην ε, πρόσβαση στα μέσα αυτά και εδώ πέρα το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβουν τα ενία και θα πρέπει να φροντίσουν ε, και η διάγνωση, η αποκατάσταση και η περίθαλψη όλων των πολιτών να είναι ιδανική. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστές στρατηγικές για την πρόληψη, για την έγκαιρη προειδοποίηση και παρέμβαση των βαρικών στα συστήματα υγειονομικής περιθάλψης και η πρόσβαση στην ε, φροντίδα είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα πρέπει να απολαμβάνουν όλοι. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία ή με το τμήμα του σώματος που έχει πρόβλημα. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες αποζημιώνονται μόνο ένα εμφύτευμα για δύο αυτιά που έχουν πρόβλημα. Ευχαριστώ. Thank you so much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενο ομιλητή είναι από την Εστονία. Βάλμαρ Άμπελ ονομάζεται. Ευχαριστώ, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ κυρίες και κύριοι από όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους Λιθουανούς γιατί εκείνοι μου ζήτησαν και μου επέτρεψαν να μιλήσω στην πανέμορφη μητρική μου γλώσσα ε, τα εσθονικά αντί να μιλήσω αγγλικά που σκόπευα αρχικά. Εκπροσωπώ ε, την εσθονική Ένωση για τη Δυσχυδή Ράχη και την Ιδροκεφαλία Αντίστοιχε οργανώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν ακόμη να εκπροσωπήσουν επάξια τους, τα μέλη τους. Για παράδειγμα, είμαστε και εμείς φορολογούμενοι και πληρώνουμε ε, τέλη συνδρομητικά, μπορούμε να ε, προσλάβουμε καλούς δικηγόρους ε, στην Εστονία τουλάχιστον και μπορούμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας στα δικαστήρια ε, να οργανώνουμε αρκετά δαπανηρές ε, μαθητείες ή σεμινάρια κατάρτισης. Αν το συγκρίνετε όμως αυτό με, τους, ε, με τις ιστονικές οργανώσεις για τα άτομα με αναπηρίες, δεν έχουν αντίστοιχα κονδύλια να προσλαμβάνουν ικανούς δικηγόρους που θα δίνουν μάχη για τους πελάτες τους. Όλα γίνονται θελοντικά και επιπρόσθετα με την κανονική απασχόληση. Δεν υπάρχει καν ε, ταμείο στην Ένωσή μας για τα δικαστικά έξοδα. Σε περίπτωση που ε, επιδιώκουμε μια δικαστική διεκδίκηση. Και έτσι κανένας δεν μας παίρνει στα σοβαρά. Στο μέτρο που οι οργανώσεις μας, οι αναπηρικές μας οργανώσεις ε, δεν θα είναι σε θέση να προσλαμβάνουν καλούς δικηγόρους, τότε τότε δεν πρόκειται το κράτος να μας λάβει σοβαρά υπόψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας θερμά και τους διοργανωτές για το πολύ ωραίο ημερολόγιο που μου χαρίσατε και που το χρειαζόμουν άλλωστε πολύ. Thank you so Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο Πίτερ Βαν Hallo, e- Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Είμαι εδώ από το EDBU, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κοφών και Τύφλων, που αποτελούν μια πάρα πολύ ευάλωτη ομάδα, η οποία συχνά, δεν ξεχνάμε, σε πολλές περιπτώσεις ε, μιλάμε για τους κοφούς, για τους τυφλούς, αλλά ε, όταν είναι κανείς και κοφός και τυφλός ε, συνδυάζει τα δύο αυτά στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να δούμε αυτή την υποτιτλισμούς. Δεν ακούμε τις περιγραφές σας. Οι λύσεις ε, για τους τυφλούς ή τους κοφούς δεν είναι λύσεις για μας. Έχουμε πολύ ξεχωριστές ανάγκες και αναγνωρίζεται η αναπηρία μας ως ιδιαίτερη αναπηρία. Χρειάζεται ειδική άμα διερμηνής. Για τους κοφούς τυφλούς ε, για την ανταλλαγή ε, εμπειρογνωμοσύνης για την βοήθεια και την εκπαίδευση τα άτομα με κόφωση και τυφλότητα και επίσης ε, δυνατότητες για χρήση ειδικών δερμηνέων προκειμένου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να συμμετάχουμε σε, στη διαδικασία προάσπιση των δικαιωμάτων μας, να ακουστεί και η δική μας η φωνή. να υπάρχουν μέσα για την ε, συμπερίληψη των κοφότυφλων. Παραν τούτον, χρειάζεται βοήθεια για την καθημερινή μας ζωή, για να μπορέσουμε να ζούμε ανεξάρτητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η πρόεδρο Ο επόμενος ομιλητή από την Ομοσπονδία Προσώπων με Αναπηρία τη Ιρλανδία, ο Γκέραντ, η Γκέραντ, πιο σωστά, Έλλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα σας μιλήσω για την τεχνολογία, αλλά όλα αυτά που λέω ισχύουν και για παιδεία μεταφορά, περιβάλλον κλπ. Θα πρέπει να είναι περίπλοκη για να είναι αποτελεσματική. Έχω ένα ρολόι Bright το οποίο το αγγίζω εδώ την ώρα και έχω εκεί πέρα και ε, διάφορα τέτοια gadget και έτσι έχω επίσης και ένα αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο και αυτό είναι προσωπικό ανάγκε μου. Παρ' όλα αυτά όμω έχουμε αναπτύξει διάφορε τεχνολογίε, ε, τι χρησιμοποιούμε για την τεχνητή ευθεία και έχουμε ε, χθε εκείνο το φόρουμ που αφορά την εικονική πραγματικότητα. Ενδιαφερόμαστε για τα γυαλιά Google, διαφορέ μηχανέ και δεν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι νέε τεχνολογίε δεν θα πρέπει να αποτελούν δεσμενή διάκριση όπω ε, είναι αυτό κάτι το οποίο θα την υπόλοιπη κοινωνία. Χρειάζεται δικαιοσύνη, δεν, χρειάζεται να υπάρχουν διακρίσεις. Θα πρέπει να βρεθούμε στην θέση του να ωφεληθούμε από αυτέ τι νέε τεχνολογίε. Όπω τα αυτοκίνητα χωρί ε, οδηγό, τα νέα υλικά, το, νέο τύπο εκτύπωσης του τρισδιάστατου. Επομένως, 65% των ε, δουλειών, των επαγγελμών θα κάνει η επόμενη γενιά δεν υπάρχουν ακόμα. Άρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες και θα πρέπει αυτές οι δουλειές να είναι προσβάσιμες για μας και για τα παιδιά μας. Και αυτές οι δουλειές θα είναι προσβάσιμες, θα είναι και ανάλογες τεχνολογίες προσβάσιμες. Επομένως, θα πρέπει η πανεπιστημιακή, ε, διάφορες πλατφόρμες, οι αναπτυξιακοί ερευνητικοί φορείς όπως το ITIL να βοηθήσουν, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αυτά να κάνουν μια προσπάθεια ούτω ώστε να έχουμε μια στεγανή νομοθετική πράξη για την προσβασιμότητα και για τα οπτικοακουστικά να αναθεωρηθεί και η οδηγία 1549 για τις δημόσιες συμβάσεις και αυτό να συνοδεύεται από αναθεώρηση της νομοθεσίας για, τα, για την χρηματοδότηση και ε, η πολιτική 2020-30 να είναι σύντονη με τη σύμβαση του ΟΗΕ θα πρέπει έτσι να αλλάξει η κοινωνία μας. Ε, θα πρέπει να γίνει πιο ευχάριστη όπως να βάζεις λίγο αλατάκι στην σούπα ή ζαχαρίτσα στο τσάι. Ε, Ευχαριστούμε. Και ο τελευταίος ομιλητής ε, του δικού μας πάνελ είναι ένας ευρωβουλευτής, ο Κρίστοφ Χέκμαν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξίστοφ Χέτμαν. Κυρίες και κύριοι, δεν επιτρέπεται άτομα με αναπηρία να μην μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα στοιχειώδη δικαιώματα του πολίτη. Και όταν σκέφτομαι τα δικαιώματα, έχω υπόψη την αξιοπρέπεια, την ανεξαρτησία, την καλύτερη προσβασιμότητα, την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και ε, βλέποντας σήμερα την κατάσταση είστε σε θέση να αξιολογήσετε καλύτερα ε, την κατάσταση. Σε μερικές χώρες έχουμε πολλές θετικές αλλαγές, αλλά έχω απόλυτη επίγνωση ότι μακρύς είναι ο δρόμος μπροστά μας ώστε πραγματικά να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες τα άτομα με αναπηρίες για να έχουν ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση. Και εμείς ε, οι εκπρόσωποι των πολιτών στα κοινωτικά θεσμικά όργανα πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά. Και χαίρομαι που ολοκληρώθηκε ήδη η πρώτη φάση των εργασιών για την ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη για την προσβασιμότητα. Θα πρέπει όμως να ε, εντείνουμε τη συνεργασία μας για την άμεση εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά πρώτα απ' όλα σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε το επίπεδο απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Και είναι κρίμα να μην αξιοποιείται στο έπακρο το τεράστιο δυναμικό αυτών των ατόμων. Ε, χρειάζονται αλλαγές με κίνητρα προς τους εργοδότες, με ενάψματα προς τους εργοδότες, με τη στήριξη στην ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, με τη θέσπιση ελαστικών ε, εργασιακών συνθηκών, με αύξηση της πρόληψης ατόμων με αναπηρία, επίσης με εξασφάλιση καλού επίπεδου ε, εκπαίδευσης προσιτή σε όλους. Σε όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αποφύγουμε ε, πολιτικές που θα διονύζουν τις διακρίσεις τα άτομα με αναπηρία που για πολλούς και διάφορους λόγους δεν ολοκληρώνουν την σπουδή, τις, τις σπουδές τους, θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να συμμετέχουν σε προγράμματα διαβίου κατάρτισης. Και τέλος, θα ήθελα να πω το εξή. Εδώ και πολύ καιρό ε, είχα να γίνω μάρτυρας τόσων χαμόγελων, τόσο, τέτοιου ενθουσιασμού σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Μας ε, περιποιείτε μεγάλη τιμή με την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρέμβασή σας και για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Ξέρω ότι πολλοί ακόμα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Είχαμε και άτομα σε λίστα αναμονής, αλλά δυστυχώς ο χρόνος πιέζει. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τα χρονικά περιθώρια και έχουμε ξεπεράσει μάλιστα και το χρονικό πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν πριν κλείσουμε το τμήμα αυτό της εκδήλωσης ε, να δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Βαρτακαστάνη. Καστάνη. Σας ευχαριστώ και ε, θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Τώρα θα προχωρήσουμε και εγκρίνουμε το ψηφίσμα. Ρώτησα την Επιτροπή προηγουμένως κατά πόσο θα ήθελε να πάρει το λόγο να σχολιάσει αυτά που παρουσιάσαμε στο ίδιο το ψήφισμα. Δύο λεπτά θα πάρει το λόγο αν το επιθυμεί για να σχολιάσει. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για άτομα με αναπηρία. ερώτηση σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα. Με τόσα πολλά άτομα που έχουν προσέλθει και η 20η επέτειος του EDF αποτελεί σημαντική ημερομηνία και καταδεικνύει ότι είσαστε μια οργάνωση με πολύ σωστή εκπροσώπηση. Μια τέτοια οργάνωση λοιπόν πρέπει να την εισακούμε. Και αυτό που θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε τη δράση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα το κάνουμε λοιπόν αυτό μόνοι μα. Έχουμε αύριο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπω σα υποσχέθηκα, θα απευθύνω έκκληση προ του υπουργού. Ελπίζω αύριο να καταλήξουμε σε συμφωνία για την πράξη, για την προσβασιμότητα, η οποία αύριο περιλαμβάνεται στην ε, η μερίσια διατάξη θα συμμετέχει και η Επίτροπος Γιούραβα και επίσης θα του παρακαλέσει να προχωρήσουν σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση για μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Δέκα χρόνια έχει κλείσει. Επιτέλους θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και θα εξετάσουμε λεπτομερώς και το κείμενο του ψηφίσματος του EDF. Να σας πω το εξή. Ε. Το γνωρίζουμε και το ακούσαμε και σήμερα ότι εσείς δεν θέλετε ακόμα λόγια, θέλετε δράση. Αλλά για να υπάρξει δράση θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, ένα πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό σήμερα που ακούσαμε το μήνυμα που α, μας δώσατε. Και να λάβουμε λοιπόν και το ψήφισμα, ελπίζω από πλευρά CDF, να υπάρχει μαζική υποστήριξη προκειμένου να το πάρουμε αυτό μαζί για την προετοιμασία της επόμενης στρατηγικής μας συνεχίζουμε την εργασία για την υλοποίηση της τρέχουσας στρατηγικής, αλλά για τα εργαλεία που έχουμε θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και για την μελλοντική στρατηγική, προκειμένου να είναι ομαλή η μετάβαση στην επόμενη περίοδο. Και διαπίστωσα λοιπόν ότι το ψήφισμα είναι πάρα πολύ ε, σύντομο, δεν περιλαμβάνει πολύ χαρτούρα. Δυόμιση σελίδες ίσα ίσα. To the point. Και κάθε σημείο λοιπόν, κάθε τέτοιο point θα το πάρουμε υπόψη στη στρατηγική μας. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο στα ωραία μας γραφεία, στο χρυσελεφάντινο πύργο μας, όχι. Συνεργαζόμαστε και με το EDF και με όλες τις οργανώσεις εξ των οποίων μιλάτε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν κύριε Βαρδακαστάνη. Νομίζω ότι με τον τρόπο σας όχι μόνο επικρίνεται, συγγνώμη, υποδέχεστε και εγκρίνεται αυτό που είπε ο Επίτροπος, αλλά εγκρίνεται το ψήφισμα, έτσι δεν είναι. Άρα, ξεκινάμε την εκστρατεία για την μέλουσα στρατηγική για τους ανθρώπους με αναπηρία. Όλα αυτά διαβιβάστε τα στους υπουργούς στη χώρα σας ολοκληρώσουμε αυτό το πάνελ και θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε όλου, όσου έλαβαν το λόγο, στου συμμετέσχων, όλοι όσοι μίλησαν και συγγνώμη σε όσους δεν προφτάσαμε να καλύψουμε. Και στο σημείο θα ήθελα να κλείσω αυτό το τρέχον πάνελ και περιμένουμε τους ε, συμμετέχοντες του επόμενου πάνελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας, όλους σας ε, και να ευχαριστήσουμε όλους ιδιαίτερα την κυρία Επίτροπο. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ λάβετε θέση για να περάσουμε στην τρίτη θεματική ενότητα της σημερινής μας διάσκεψης. And if you do so, then I will use the excellent opportunity σκοπεύω να αξιοποιήσω αυτή την εξαιρετική ευκαιρία που μας δίνεται να μιλούμε τη μητρική μας γλώσσα και εγώ θα μιλήσω τα τσεχικά που είναι η μητρική μου γλώσσα. Αξιότιμα μέλη εκπρόσωποι των οργανώσεων, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, με τιμά ιδιαίτερα ε, η δυνατότητα που έχω να προεδρεύσω σε αυτό το τρίτο τμήμα της εξαιρετικής αυτής σημερινής εκδήλωσης. Ονομάζομαι Όλγα Σεχνάλοβα και είμαι Ευρωβουλευτής από την Τσεχία στο κόμμα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και είμαι συμπρόεδρος της ε, Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με αναπηρίες. Συνεδριάζουμε σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρά του γεγονότος αυτό ή μάλλον ακριβώς εξαιτία αυτού του γεγονότος δεν θα πρέπει να μιλούμε μόνο για τα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θυμηθούμε τα 800 δισεκατομμύρια ατόμων με αναπηρία ανά την υφήλιο, που μερικές φορές είναι τελείως απομονωμένα και στο περιθώριο της κοινωνίας. Και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν πρόσβαση σε παιδεία, στην υγεία και σχεδόν είναι αδύνατο να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Η αναπηρία είναι από τους βασικότερους στόχους, ε, από τις βασικότερες αιτίες της φτώχειας ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε την υλοποίηση του 17ου βιώσιμου αναπτυξιακού στόχου, που είναι η εξάλληψη της φτώχειας με κάθε μορφή στον κόσμο ολόκληρο. Και βασικός ε, στόχος των βιώσιμων στόχων της ανάπτυξης των ΗΕ Εθνών είναι να μην αφήσουν κανέναν πίσω, να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των πολιτών και να συμπεριλάβουν και το άτομα με αναπηρία σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και σε όλες τις σφαίρες δραστηριότητες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να λάβουμε λοιπόν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να τις ικανοποιήσουμε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα άτομα αυτά στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και μάλιστα σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της θέσπισης αλλά και της ε, εφαρμογής. Με ιδιαίτερη χαρά θα συμπροεδρεύσω ε, μαζί με την Άντια Χαντάντ, μέλος της ε, Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Θα προεδρεύσουμε θα συμπροεδρεύσουμε σε αυτό το τρίτο σκέλος της διάσκεψης. Επειδή έχουμε ήδη μείνει πίσω, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξάλεπτο που έχετε για τις παρουσιάσεις σας. Πρώτα θα μας μιλήσει ο Επίτροπος Νέβεν Μίμιτσα, αλλά από βίντεο. Παρακαλώ, θα ακούσουμε τον Επίτροπο Μίμιτσα. Κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, ε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά εκφωνώ ομιλία σε αυτό το τέταρτο Ευρωκοινοβούλιο των ατόμων με αναπηρία. Το φετινό Ευρωκοινοβούλιο συμπίπτει με την 20η επέτειο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Τα τελευταία 20 χρόνια έχετε τιμήσει το σύνθημά σας. Τίποτα για μας χωρίς εμάς. Με το δικό σας έργο και προσπάθεια εξασφαλίζεται ισχυρή και θετική εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βοηθάτε καθημερινά να διαμορφώσουμε μια πιο συμμετοχική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με ίσες ευκαιρίες για όλους. Μαζί σας λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον κόσμο. Όπως ξέρετε, διαδραματίσαμε κέριο ρόλο ζητώντας υψηλότερες φιλοδοξίες από το νέο Παγκόσμιο Θεματολόγιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 με την υπόσχεση να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Για πρώτη φορά αυτό το νέο παγκόσμιο πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές στα άτομα με αναπηρία. Αυτό ήταν κάτι το ρηξικέλευτο για το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους στο, στον κόσμο που βιώνουν κάποιο είδος αναπηρίας. 80% αυτών των ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση είναι πλήρε συμβαλόμενο μέρο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ω περιφερειακή οργάνωση. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει και την ειδική δέσμευση να μεριμνήσει για μια διεθνή συνεργασία που θα είναι συμμετοχική και προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρίες. Το 2015 τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν τη θετική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως προς την εφαρμογή της σύμβασης, ιδιαίτερα κατά τη χρηματοδότηση των εξωτερικών μας δράσεων. Φέτος το καλοκαίρι όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και 28 χώρες μέλη υιοθέτησαν ένα νέο, μια νέα ευρωπαϊκή συνένεση για την ανάπτυξη. Η νέα αυτή συνένεση εδράζεται στα υπάρχοντα πλαίσια πολιτικής για τις αναπηρίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και διατρανώνει τη δέσμευσή μας για μια δικαιωματική προσέγγιση της ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας το σύνδεσμο μεταξύ φτώχειας και αναπηρίας. Επίσης, η συνένεση αυτή αναφέρεται ρητά στα άτομα με αναπηρία, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να λάβει υπόψη τις ειδικέ τους ανάγκες και να εξασφαλίσει την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Βέβαια, δεν δίνουμε απλώς το καλό παράδειγμα με τα λόγια μας, αλλά το δίνουμε και με τα έργα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός δωρητής που στηρίζει τα δικαιώματα και την εσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία παντού στον κόσμο. Και από το 2010 έχουμε χρηματοδοτήσει πάνω από 330 ειδικά σχέδια για την αναπηρία σε πάνω από 95 χώρε σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προωθώντα τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στην, στην Αφρική, βελτιώνουν την πρόσβαση στην σωματική αποκατάσταση στο Αφγανιστάν ή ε, δίνοντας σε νεαρούς κοφούς ε, την πρόσβαση στην πληροφορία ε, για σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα στην Παραγουάη και την Ουρουάη. Και αυτά είναι μόνο λίγα παραδείγματα των δράσεών μας. Πρόσφατα μάλιστα εγκαινιάσαμε δύο συγκεκριμένες δράσεις για να συνεκτιμήσουμε την ε, διάσταση της αναπηρίας στους διαλόγους μας για την πολιτική και τις παρεμβάσεις μας στις χώρες εταίρους. Μόλις χθες εγκαινιάσαμε ένα τετραετές πρόγραμμα με τίτλο «Γεφυρώνοντας το χάσμα» προκειμένου να ε, βοηθήσουμε για την εφαρμογή συμμετοχικών πολιτικών και υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμού στα άτομα με αναπηρίες. Το θέμα μάλιστα Τη φετινή διεθνού ημέρα για την αναπηρία είναι η μεταμόρφωση, ο μετασχηματισμό προ μια βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία για όλου. Και μάλιστα η Γεντνεμπέρ Σνιγκούση, μια επιφανής ε, υπέρμαχο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ε, Αιθιοπία, ενσαρκώνει ακριβώ αυτού του είδου τη μεταμόρφωση. Γιατί βοηθώντα του άλλου με κίνητρο τη διακρίση που υπέστη ίδια ως νέα ε, τυφλή Αφρικανή, μα υπενθυμίζει ότι η ηγετική ικανότητα δεν συνδέεται ούτε με τα μάτια μα ούτε με τα αυτιά μα ούτε με τα πόδια μας. Πηγάζει όμως από μέσα μας και ο καθένας από μας έχει την ικανότητα να γίνει ηγέτης όπου και αν βρίσκεται και έχει την ικανότητα να βοηθήσει τους γύρω του να διάγουν μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να κατακλείδει να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ηγέτες που βρίσκονται εδώ σήμερα στην αίθουσα γιατί μας βοηθούν να μην αφήσουμε πραγματικά κανέναν πίσω προσβλέπω σε στενή συνεργασία μεταξύ μας ώστε να προωθήσουμε τα δικαιώματα και την εσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία παντού στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, nyní je mi Σας ευχαριστούμε εμείς, λέει η Πρόεδρος. Και με ιδιαίτερη χαρά που δεχόμεθα τον Χρήστο Στυλιανίδη, τον Επίτροπο με το χαρτοφυλάκιο της ανθρωπιστικής ε, βοηθείας και διαχείρισης των κρίσεων. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε Βαρδακαστάνη, λέει ο κύριος Τηλιανίδης, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, για μένα αποτελεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση να είμαι σήμερα εδώ σε αυτή την σημαντική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Προσώπων με Αναπηρία ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους. Έτσι μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις στο σημαντικό σας φόρουμ. Μόλις πριν από λίγες μέρες γιορτάσαμε την Ευρωπαϊκή Μέρα προς τιμή των προσώπων με αναπηρία. Πρόεδρε Παρατακαστάνη, επιτρέψτε μου να στείλω τις καλύτερες ευχές μου για την 20η επέτειο τις δράσεις του Ευρωπαϊκού σας φόρουμ. Και γνωρίζετε καλύτερα από μένα κυρίες και κύριοι ότι υπολογίζουμε σε ένα δισεκατομμύριο α, τους ανθρώπους με αναπηρία. Και το 80% από αυτούς βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Δυστυχώς. Ακόμα και στις ανεπτυγμένες χώρες οι άνθρωποι με αναπηρία πολύ συχνά μειονεκτούν στην κοινότητα όπου ζουν. Ε, βέβαια, στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες έχουν πιο πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίζουν περισσότερες δεσμενείς διακρίσεις. Ακόμα και σε περίοδο που δεν σοβεί κάποια κρίση στην χώρα τους. Παρ' όλα αυτά, οι εκτοπισμοί ε, και οι θεομηνίες πίσω αυτές τις χώρες, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε βοήθεια και σε αρρωγή. Γίνεται όμως πιο δύσκολη άρα χρειάζεται περισσότερη προστασία για τις βασικές υπηρεσίες. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί περιορισμοί και η βοήθεια δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Τρόφιμα, νερό, υγιεινή. Πάντως, πολλές φορές και που είναι πιο σημαντικό, χρειάζονται και ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Πολύ συχνά. Άνθρωποι με αναπηρίες μένουν στο περιθώριο. Δεν λαμβάνουν υπόψη από τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και από την ανάπτυξη αυτών. Και από την Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι και διαμορφώνουμε το παγκόσμιο ανθρωπιστικό πλαίσιο και περιβάλλον. Την περασμένη εβδομάδα, περασμένη χρονιά μάλλον, φτάσαμε στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σαφής η εντολή μας και η δική μου εντολή ως Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση των κρίσεων. Πρέπει να βοηθούμε τους πλέον ευάλωτους. Και οι άνθρωποι με αναπηρίες θα πρέπει να είναι κορυφαία μας προτεραιότητα. Είναι ηθικό μας καθήκον ως Ευρωπαίων. Είναι ε, πολύ σημαντικό ρόλο τη Ένωση για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων αυτών. Πρώτον, εμεί έχουμε προσχωρήσει στην ε, σύμβαση του ΟΗΕ για τα πρόσωπα με αναπηρία και αυτό καλύπτει και προβλέπει συγκεκριμένε υποχρεώσει μα σύμφωνα με το άρθρο 11, ιδίω όσον αφορά κάποια κατάσταση κρίση και κάποιε ε, κατεπίγουσε καταστάσει. Οπότε θα πρέπει αυτέ οι υποχρεώσει να αντικατοπτρίζονται στις πολιτικέ μα. Για κάθε πτυχή του. Δεύτερον, έχουμε εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης για όλες τις ε, ε, πρακτικές πλευρές της δέσμευσής μας, της διεθνούς. Όμως, το θέμα δεν είναι μόνο τα λόγια. Χρειάζονται και συγκεκριμένες πράξεις. Πρώτα-πρώτα, ενσωματώσαμε τις ανάγκες αυτών των ε, προσώπων στις πολιτικές μας. Προστασία, αναγκαστική ε, εκτοπισμό και επίσης όσον αφορά τα, της υγείας και υγιεινής. Φέτος δεν χρηματοδοτούμε τις κατευθυντήριε γραμμές για πρώτη φορά για να καλύψουμε και τα πρόσωπα με αναπηρία στην ανθρωπιστική δράση. Έτσι αποδεικνύεται η δέσμευσή μας να αλλάξουμε το σύστημα σε κάθε πλευρά του. Επίσης, δίνουμε στοχισμένη χρηματοδότηση για συγκεκριμένη βοήθεια σε, ε, που έχουν αναπηρία εκεί όπου έχουμε κάποιου είδου ε, θεομηνίες και κρίσεις. Τα πρόσφατα χρόνια είχαμε 26 τέτοια προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και διαθέσαμε 30 εκατομμύρια ευρώ. Και από την αρχή της εντολής μου αύξησα αυτή την χρηματοδότηση κατά 40% και πάνω. Μερικά παραδείγματα για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε που ανέλαβε αυτό το ε, χαρτοφυλάκιο στην Τουρκία. Βελτιώσαμε την ε, πρόσβαση σε επιδικές υπηρεσίες για τους πρόσφυγες που έχουν κάποια αναφερία. Στο Νότιο Σουδάν βοηθήσαμε ούτως ώστε να υπάρξει δημιουργία δυνατοτήτων των ε, παραγόντων ανθρωπιστική βοήθεια και έτσι να εξασφαλίσουμε την κάλυψη των προσώπων με αναπηρία. Στην Ινδία χρηματοδοτήσαμε την πρόσβαση σε αποκατάσταση σωματικών προβλημάτων των προσώπων με αναπηρία. Στη ΔΕ Ελλάδα χρηματοδοτήσαμε την δημιουργία κάποιων καταφυγίων στέγασης ε, τέτοιων προσώπων και επίσης την παροχή των διατροφής. Και συνεχώς προβληματιζόμαστε, συζητούμε πώς μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερο με τους συνομιλητές μας που δρούν επί τόπου. Επίσης, πετύχαμε πάρα πολλά όσον αφορά την ε, πολιτική προστασία και το πώς εκεί θα έχουμε ένταξη που και αυτό είναι θέμα του χαρτοφυλακίου μου και έτσι στην διαχείριση των ε, θεομηνιών καλύπτουμε και τους ανθρώπους με αναπηρία, ετοιμάζουμε κάποια προγράμματα για αυτούς που πάσχουν κάποια αναπηρία. Προ δύο ετών δε το Συμβούλιο ενέκρινε τα σχετικά συμπεράσματα όσον αφορά τη διαχείριση των ε, θεομηνίων ε, για να καλύψουμε και τις συγκεκριμένες ανάγκες των όσων έχουν κάποια αναπηρία. Πολλά κάνουμε, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα Όλοι μαζί. Οι δύο ιδιοσυντορητές, οι εταίροι μας και είμαι έτοιμος ως Επιτροπός να αναλάβω περαιτέρω δράση τόσο ώστε να μπορέσω να καλύψω τις ανάγκες όσων έχουν αναπηρία και αυτό να γίνεται επιτόπου και παντού. Αγαπητοί φίλοι, καμιά φορά μου λένε ότι θα πρέπει πρώτα να έχουμε μια κοινωνία που να είναι φιλική προς τους με Πριν όμως φτάσουμε σε αυτή τη φάση, να δούμε τι γίνεται με τις κρίσεις. Και νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι κοντόφερμα. Βέβαια και έχουμε διάφορα προβλήματα να λύσουμε στην Ευρώπη, στις χώρες μας. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας σταματά από το να προσπαθούμε να υπάρχει κάποια ανθρωπιστική δράση που να ενσωματώνει περισσότερο. Η μία προσπάθεια δεν ακυρώνει την άλλη. Και τα δύο αυτά μέτωπα ε, συγκλίνουν και το ένα ενισχύει τις προσπάθειες για το άλλο. Τους πρόσφατους μήνες συζήτησα με φορείς προσώπων με αναπηρία για να δούμε με τους εταίρους μας πώς μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων και η σχετική δέσμευση είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε. Και πριν από λίγε μέρε είχα τη χαρά να δω τον πρόεδρο Βαρδακαστάνη και συμφωνήσαμε όσον αφορά το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία που να ενσωματώνει περισσότερο παντού. Και όπως ε, είπαμε, είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να καταφέρουμε περισσότερα. Και έτσι θα καταφέρουμε τα περισσότερα. Πρώτα-πρώτα, για πρώτη φορά η χρηματοδότησή μας που εξαγγελθήκε αποδεικνύει ότι θα πρέπει οι εταίροι μας να καλύψουν ε, τους ανθρώπους με αναπηρία στις σχετικές δράσεις. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερον, πρόκειται να επεξεργαστούμε κάποια πρότυπα για την ανθρωπιστική δράση της Ένωσης και έτσι συγκεκριμένες ανάγκες των ευάλωτων ομάδων όπως ανήλικοι ή παιδιά με αναπηρία επαρκώς θα καλυφθούν. Τρίτον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα πρόσωπα με αναπηρία είναι εις θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους και αυτές να λαμβάνονται υπόψη συνέχεια όχι μόνο όταν είναι αποδέκτες ανθρωπιστικής δράσης, αλλά και ως ε, ενεργοί ε, συνεργάτες στην λήψη των σχετικών αποφάσεων. Αυτό είναι προσωπική μου δέσμευση. Ε, τα πρόσωπα με αναπηρία να είναι συνομιλητές μας διαβούλευση για κάθε πρωτοφουλία μέσω των φορέων που τους εκπροσωπούν. Ε, είμαστε εμείς προσιλωμένοι στο ότι τίποτε για τους ανθρώπους με αναπηρία δεν πρέπει να αποφασίζεται χωρίς την συμμετοχή αυτών στις αποφάσεις. Πέρσι χρηματοδοτήσαμε ένα στεγανό γερό πρόγραμμα στην Μιανμάρ και πρόσωπα με αναπηρία επίσης είχαν εμπλακεί όσον αφορά την πρόληψη, την, την περιστολή των καταστροφών και του είπε κάποια σοφά λόγια κάποιος ότι εάν έρθει κάποια καταστροφή ε, τότε όλοι θίγονται. Οπότε και όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν όσον αφορά την προπαρασκευή μας για τις καταστροφές αυτές. Αν θα πρέπει να δούμε το πώς θα μπορούμε να καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπους με αναπηρία στα όσα κάνουμε. Να έχουμε καλύτερη συλλογή δεδομένων. Και τελευταίο αλλά σημαντικό, θα πρέπει να προσυλλοθούμε στη δημιουργία δυνατοτήτων για το πώς θα δουλέψουμε επίσης προς το να υπάρχει μεγαλύτερη ένταξη των προσώπων με αναπηρία και πώς η γνώση θα γίνει κοινό κτήμα και πώς ε, επίσης θα ενισχύσουμε την εκπροσώπηση. Πριν από λίγε μέρε, αγαπητοί φίλοι, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε μια έκθεση που αφορούσε την εφαρμογή, την υλοποίηση τη στρατηγική για του ανθρώπου με αναπηρία. Και λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν θα πρέπει να μείνουν πίσω. Δεν θα πρέπει να μένουν, μείνουν έξω από την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. Και συμφωνώ 100% γιατί είναι αυτό καθήκον μα. Και πάντοτε είμαι έτοιμο να ακούσω τι δικέ σα προτάσει για να βελτιώσουμε το τι κάνουμε με τους ανθρώπους με αναπηρία και κυρίως όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Δυστυχώς μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Πρόκειται για μια διαδρομή, μια διαδικασία που απαιτεί συλλογική δράση Ο πλευρά όλων. Όμως είναι κοινό συμφέρον μας να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτο σε περίπτωση κρίσης. Νομίζω ότι μαζί αυτή η αρρωγή μπορεί να καλύψει περισσότερους και μαζί μπορούμε να κάνουμε την διαφορά όσον αφορά τις ζωές των ευάλωτων. Πιστεύω ότι χέρι-χέρι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Commissioner. Σας ευχαριστώ, Επιτρόπε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ συγκεκριμένη, στοχευμένη και ενημερωτική σας παρέμβαση. Νομίζω ότι όλες, όλοι μας το εκτιμήσαμε. Και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Γιώζεπ Μαριά Τερικάμπρας, αντιπρόεδρο των Πρασίνων και EFA, μέλος τη ε, κοινή ε, κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικό και Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιπροσωπεία στο Μεξικό. Ναι, σας ζητώ συγγνώμη, θα είμαι συντομό γιατί θα πρέπει να φύγω μετά την σύντομη παρέμβαση μου. Έχω διαφορετική μια άλλη συνεδρίαση να παρευρεθώ. Σα ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι αγαπητοί φίλοι, είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να απευθύνω το λόγο σε εσά και εξ ονόματο του κυρίου Φίλιπ Λάμπερτ, συμπρόεδρο τη ομάδα αυτή στο Κοινοβουλίο. Η ομάδα μας πάντα προασπιζόταν την ίση αντιμετώπιση για τα άτομα με αναπηρία και θα συνεχίσει, θα συνεχίσει να το πράττει σε όλα τα επίπεδα. Με προτεραιότητα στην προσβατιμότητα, την προσβατιμότητα στη συμμετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, υγεία, κοινωνική προστασία και εξωτερική δράση. Στι 30 Νοεμβρίου φέτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς περάσαμε ένα ψήφισμα για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγική για την ε, ε, αναπηρία. Εμείς λοιπόν ψηφίσαμε, η ομάδα μας ψήφισε υπέρ τη στρατηγική παρά το γεγονό ότι κάποια στοιχεία και κάποιε πτυχέ δεν συμπεριλήφθηκαν στο ψήφισμα, κυρίω ε, η αναφορά της ανατροπής της πολιτικής λιτότητος και για να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε σεξουαλικές και αναπαραγωγικές υπηρεσίες για γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία και να ανασταλούν κάποιες πρακτικές στήρωσης. Επιτρέψτε μου τώρα να πω δύο λόγια πέρα από τα συγκεκριμένα μέτρα για να κοιτάξουμε βαθιές ε, πεπιθήσεις μας. Υπάρχει η εξής πεποίθηση όλα τα ανθρώπινα όντα είναι ίσα σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι διαφορές μεταξύ μας δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση αυτή τη βασική θεμελιώδη αξιοπρέπεια. Έτσι περαιτέρω, αν κάποιος ε, εκ λόγω ατυχήματο ή λόγω άλλων συνθήκων έχει αναπηρία, δικαιούται να λαμβάνει υποστήριξη και βοήθεια από την κοινωνία και δικαιούται να συναποφασίζει για τα ποια είναι τα καλύτερα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό επειδή είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά, είμαστε ανθρώπινα όντα, ανθρώπινα όντα με μια ζωή η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί, να προοδεύσει, να εξελιχθεί με προσδοκίες, με συναισθήματα, με ανάγκες, με φόβους και ελπίδες. Η υποστήριξή μας λοιπόν στα άτομα με αναπηρία δεν αποτελεί μία σύμβαση από αυτούς που δεν έχουν αναπηρία. Όχι, είναι αναγνώριση της κοινή μας επιθυμίας, της κοινή μας μοίρας αυτή τη γη. Γι' αυτό η συμμετοχή σας και η συνεργασία σας χρειάζεται ανα πάσα στιγμή, στα πάντα, σε ό,τι κάνουμε για κλάδους τους οποίους γνωρίζετε πολύ καλύτερα από ότι εμείς. Να είσαστε βέβαιοι για το εξή. Μπορείτε να υπολογίζετε στη μόνιμη αλληλεγγύη μας, όπως ζητάμε αλληλεγγύη από όλους όσοι πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο να ζήσει κανείς σε ένα καλύτερο κόσμο, να ζει κανεί σε ένα κόσμο που σέβεται τις ανθρώπινες αξίες και την αξιοπρέπεια όλων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, για την κατανόησή σας, ακόμα και όταν δεν είμαστε τόσο δραστήριοι όσο θα έπρεπε να είμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ιωζεπ. Κυρίες και κύριοι, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και εφαρμογή τους ε, είναι ένα θέμα που το παρακολουθεί εκ του σύνεγγης ε, η SDG Watch Europe και καλωσορίζω την πρόεδρο Άλισο Κόλμαν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση της SDG Watch Europe για να λάβουμε μέρος στη συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Επίσης να πω χρόνια πολλά στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων ε, με αναπηρία που συμπλήρωσε τα 20 χρόνια Λέγομαι Άρισον Κόλμαν. Ε, είμαι στην ε, Διεθνή Διαφάνεια για θέματα πάταξης διαφθοράς ε, και στον ελεύθερο μου χρόνο συμμετέχω και στην SDG Watch. Εδώ εκπροσωπώ την SDG Watch. Καταρχήν να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας για το τι σημαίνει η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί ήταν περίπλοκη η διαδικασία. Αυτό που είναι η στόχη αυτή, η βιώσιμης ανάπτυξη, είναι μοναδικής σημασίας πολιτική δέσμευση και ζητούν καινοτόμε δράσει από όλε τι χώρε για την ευημερία και την προστασία του πλανήτη. Καλύπτουν οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα διακυβέρνηση. Την υγεία, την κοινωνική προστασία, την παιδεία, τις, την απασχόληση, τι κλιματικέ αλλαγέ, την περιβαλλοντική προστασία, τη δικαιοσύνη και του ισχυρού θεσμού. Αυτή η 17 στόχη είναι η αναγνώριση ότι μόνο χάρη στενή συνεργασία σε όλους αυτούς τους τομείς μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές. Και αυτή η ευρεία προσέγγιση δεν είναι το μόνο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των στόχων αυτών. Η ενσωμάτωση βρίσκεται στην καρδιά του, στο επίκεντρό του, δηλαδή η χειραφέτηση, η αποφυγή των διακρίσεων. Εξού και το σύνθημα να μην μείνει κανένα πίσω και το όραμα μια δίκαιη, ανοιχτή, ανεκτική, περιεκτική, συμμετοχική κοινωνία χωρί αποκλεισμού, με λήψη υπόψη τη ανάγκη των πιο ευάλωτων. Κάθε χώρα στον κόσμο, είτε είναι αναπτυσσόμενη, είτε αναπτυγμένη, είτε είναι εύπορη, είτε φτωχή, κάθε χώρα του κόσμου έχει ε, ευθύνη να κατευθύνει τι πράξεις και τι ενέργειές τη υπέρ τη υλοποίηση των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη και όλοι θα πρέπει να δεσμευτούν ε, να υλοποιήσουν τους 17 στόχους και τους 169 σκοπούς ε, και να μην ξεχνούμε τις πιο ευάλωτες ομάδες ε, των συμπολιτών μας. Δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί ηγετική ικανότητα και φυσικά πολύ σκληρή δουλειά. Και κάτι τέτοιο θα σημαίνει αναζήτηση νέων τρόπων εργασίας, νέων τρόπων σκέψης και οπωσδήποτε θα πρέπει να βρούμε και νέους τρόπους συνεργασίας. Και αυτό ακριβώ κάνει η ομάδα μας, η SDG Watch Europe, που ε, έχει συμπληρώσει μόλις τα δύο χρόνια και ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2015. Είμαστε ένα δίκτυο οργανώσεων με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Πάντω, συνεργαζόμαστε για την εφαρμογή των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να φέρουμε ε, την κοινωνία των πολιτών ε, κοντά σε θέματα όπως είναι ανάπτυξη περιβάλλων ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά, άτομα με αναπηρίες, στέγαση, δικαιοεμπόριο, πάταξη της διαφθοράς, διαφάνεια. Προσπαθούμε όλα αυτά τα θέματα να τα συνδυάσουμε και όλες αυτές τις ομάδες να τις φέρουμε σε ένα κοινό τραπέζι. Έχουμε πάνω από 180 μέλη. Μερικά βρίσκονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλα σε εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μαζί από κοινού. Έχουμε συζητήσει με πολιτικού ηθήνοντε. προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε του πολίτε και παρακολουθούμε το βαθμό εφαρμογή των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της πρόοδο προ την εφαρμογή ε, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξη. Είχαμε στο πάνελ και τον αρμόδιο επίτροπο ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ θα σα ε, πω για το τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εντό τη Ευρωπαϊκή Επικράτεια, στα κράτη-μέλη. Πέρυσι είχαμε την πρώτη έκθεση για την Ευρωπαϊκή Δράση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Και παρά την υπόσχεση για την υλοποίηση των στόχων, λίγα συγκεκριμένα μέτρα υπήρχαν. Το έγγραφο εξέτασε μόνο οι φυστάμενες πολιτικές και δεν έκανε αξιολόγηση των κενών. Θα πρέπει να δούμε όμω τι αδυναμίε, τα κενά, τι λείπει, τι δεν κάνουμε ώστε πραγματικά να ε, χαράξουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια γενική στρατηγική για να προωθήσει την πολιτική συνοχή και το συντονισμό. Και αυτό θα πρέπει να το κάνει με την ενεργό συμμετοχή και ανάμειξη και των ατόμων με αναπηρία και όλων των άλλων ομάδων με κίνδυνο περιθωριοποίησης. Θέλουμε ξεκάθαρο σχέδιο εφαρμογής με στόχους και χρονοδιάγραμμα Χωρίς κάτι τέτοιο, πώς είναι δυνατόν να ε, ευελπιστούμε στο ότι θα υλοποιήσουμε ουσιαστική πρόοδο την επόμενη δωδεκαετία. Αυτή η έλλειψη φιλοδοξίας ε, που χαρακτηρίζει την πρώτη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, απόδειξη ότι η παρούσα ηγεσία δεν έχει πραγματική προτεραιότητα του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο στην ομιλία του το Σεπτέμβριο για την κατάσταση της Ένωσης δεν αναφέρθηκε ο πρόεδρος Γιουνκέρ ούτε στην ανάπτυξη ούτε στη βιώσιμη ανάπτυξη. Κάτι που δείχνει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν εμπίπτει σε αυτές τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε και πέντε σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης. Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης σε αυτό το έγγραφο των πέντε σενάριων σχεδόν δεν αναφερόταν η βιώσιμη ανάπτυξη. Απλώ αναφέρθηκε ο ηγετικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην υιοθέτηση των στόχων. Αλλά ουδή λόγο για το πώ μπορεί να ηγηθεί τη εφαρμογή των στόχων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ χάσαμε μια ευκαιρία. Γιατί οι στόχοι δίνουν ένα θετικό όραμα για την Ευρώπη. Ένα όραμα για ένα ευρωπαϊκό μέλλον που θα στηρίζεται σε αξίε. Ένα όραμα που θα ε, διασκεδάζει τις ανησυχίες όλων των Ευρωπαίων πολιτών και των πιο ευάλωτων και μειονεκτικών ομάδων και θα εξασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον. Η οργάνωσή μας, η SDG Watch και άλλες οργανώσεις έγραψαν το δικό του σενάριο, το έκτο σενάριο για το μέλλον της Ευρώπης. Με καλό σχέδιο, με σωστούς στόχους, αλλά χωρίς εργαλεία για την καταμέτρηση της πρόοδου δεν θα πάμε πολύ μακριά. Και μάλιστα η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ε, εκπώνησε την πρώτη έκθεση σε ό,τι αφορά τους στόχους με 100 περίπου δείκτες. Χαιρετίζουμε την έκθεση της Eurostat, αλλά ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Η διαδικασία της επιλογής των, 10, ε, των 100 δικτών ήταν κάπως ε, βεβαιασμένη, σπευσμένη και με λίγη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους. Η έκθεση δεν δείχνει επαρκή πρόοδο και την αποτυχία στην υλοποίηση των στόχων. Επίσης δεν καλύπτει όλες τις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης ούτε εντοπίζει τα κενά και που υπάρχουν ελλείψεις. Η έκθεση δεν δείχνει πόσο μακριά και πόσο γρήγορα θα πρέπει να κινηθούμε αν θέλουμε πραγματικά μέσα σε 12 χρόνια να υλοποιήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Λείπουν και κάποια βασικά στοιχεία από την έκθεση σε ό,τι αφορά την αρχή του να μην αφήσουμε κανένα πίσω. Δεν καταμετρά σωστά τις ανισότητες ε, ή τη μείωση των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι στόχοι υποτίθεται ότι εξυπηρετούν περισσότερο τους φτωχότερου συμπολίτε. Ε, φτωχότερους ε, Θέλουμε όμως και τοπικά ε, μεμονωμένα στοιχεία και όχι συγκεντρωτικά για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα και την πρόοδο σε επιμέρους τομείς. Πάντως, στην πρώτη αυτή έκθεση, η Ευρωπαϊκή Στρατιστική Υπηρεσία δεν συμπεριέλαβε κάποια κρίσιμα στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία για τα άτομα με αναπηρίες σε ό,τι αφορά το στόχο 4 στην έκθεση της Eurostat για την ποιότητα της παιδείας. Δεν υπήρχαν στοιχεία για τα άτομα με αναπηρίες σε ό,τι αφορά τον στόχο 8, την αξιοπρεπή απασχόληση για όλους του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρήσει το κατάλογο αυτό με τους δείκτες και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την αξιολόγησή της σε κατάλληλες και συμμετοχικές διαδικασίες. Θα πρέπει να διευρύνει τις εκθέσεις παρακολούθησης και να μην στηρίζεται μόνο σε ποσοτικούς αλλά και σε ποιοτικού δείκτες. Επίσης θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τους στόχους της στο γενι... στη γενική δέσμη στόχων και να είναι ακόμη πιο φιλόδοξη αν πραγματικά θέλει να δείξει πρωτοπορία. Επίσης, να προτείνει νέα ξεχωριστά στοιχεία που να περιλαμβάνει και ομάδες όπω άτομα με αναπηρία Να μην είναι όλα τα στοιχεία συγκεντρωτικά. Και όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να γίνουν με ανάμειξη τη κοινωνία των πολιτών. Τούτου λεχθέντος ε, ε, να καταλήξω σε ένα πιο θετικό τόνο, γιατί μέχρι στιγμή σα τα είπα κάπως απεσιόδοξα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε γενέθλια και σε κάθε γενέθλια κάνουμε ευχές για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στήσει μια πλατφόρμα με πολλούς ενδιαφερόμενους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν η κοινωνία των πολιτών, εμπειρογνώμονες, επιχειρήσεις, ε, συνδικάτα. Όλοι συνεργάζονται υπέρ της εφαρμογής των στόχων. Χθες είχαμε την πρώτη συνεδρία σε αυτή της πλατφόρμας και ήταν αρκετά ενθαρρυντική. Πραγματικά νιώθω αισιόδοξη για το μέλλον. Η πλατφόρμα αυτή θα δώσει ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καλύτερες διαβουλεύσεις και στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και άλλους εμπειρογνώμονες. Η πλατφόρμα αυτή θα δημιουργήσει μικρότερες, πιο λιγομελείς ομάδες εργασίας που θα εγκύπτουν ε, πιο εμβριθώ σε κάποια θέματα. Και πολύ πιθανόν να έχουμε και μια μικρή ομάδα για το μέλλον του κοινοτικού προπολογισμού, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώ και την αξιολόγηση και την παρακολούθηση. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει περισσότερου ενδιαφερόμενου σε αυτέ τι μικρέ ομάδε, γιατί οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν τι γνώσει του και την εμπειρογνωμοσύνη του. Και ένα από αυτού του ενδιαφερόμενου είναι και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Θα πρέπει τώρα να δείξει ηγετική ικανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή των στόχων γιατί μόνο με συνεργασία στην εφαρμογή θα υλοποιήσουμε πραγματικά ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ και κλείνοντας λοιπόν το πάνελ θα ήθελα να καλωσορίσω τον, την Αντιπρόεδρο του ETF, την κυρία Άννα Πελάε η οποία επίσης προεδρεύεται τη Επιτροπή Γυναικών στο EDF και εστιάζεται κυρίω σε θέματα ε, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η κυρία Πελάη. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τα ισπανικά. Αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ανθρώπων με Αναπηρία, αγαπητή, συνάδελφοι εδώ στο πάντως στο Προεδρείο, αγαπητοί ευρωβουλευτές, αγαπητές αδερφές και αδελφοί στην αναπηρία, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τρία θέματα. Πρώτα πρώτα, πόσο σημαντική είναι η υπόθεση θεματολογία 2020-30 και η βιώσιμη ανάπτυξη για μας τα πρόσωπα με αναπηρία. Πρόκειται για ένα αυθεντικό όραμα που έχουμε για το μέλλον, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ανθρώπινη ανάπτυξη. Και το σλόγγαν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανείς, κανείς να μην μείνει απ' έξω. Να μην χάσει το τρένο. Και ε, λόγω του κινήματός μας καταφέραμε, φίλοι, το να καλυφθούν και τα πρόσωπα με αναπηρία σε αυτή την θεματολογία της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, έχουμε τον στόχο 4 και μιλούμε για ισότητα στην εκπαίδευση. Στο 8 και που μιλάμε για αξιοπρεπή εργασία και όσο εκεί που μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη. Στο στόχο 10, εκεί που αναφερόμαστε στην ε, συρρήκνωση, στη μείωση, καταπολέμηση της ανισότητας. Και επίσης και στο στόχο 11, εκεί που αναφερόμαστε στις ε, βιώσιμες πόλεις, βιώσιμες κοινότητες, αλλά επίσης καλυπτόμαστε και στο 17, εκεί που μιλούμε για αυτή τη συμμαχία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και επίση στον στόχο 17 αποκτούμε την δυνατότητα να περνάει ε, το πρόβλημά μας και σε άλλους σημαντικούς στόχους που είναι πολύ σημαντικοί για μας άντρες και γυναίκες που έχουμε πια αναπηρία όπως ας πούμε ο στόχος 1 που είναι η καταγνώριση της φτώχειας στόχο στόχος 2 ε, τέλος στην, στην πείνα, στο λαιμό, στον στόχο 3 υγεία και ευημερία και επίσης και στο στόχο 5 που είναι η ισότητα ανδρών και γυναικών. Πόσο πραγματικά σημαντικό είναι να λαμβάνετε υπόψη το τι χρειαζόμαστε εμείς που έχουμε αναπηρία, το, το κίνημά μας και έτσι έχουμε το θεματολόγιο 2030 για αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία ούτω ώστε να μπορέσουμε ε, να έχουμε και την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία να καλυφθούν και αυτά που και αυτό είναι ε, το περιεχόμενο της δικής μας ε, πολιτικής ε, ατζέντα και τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη είχαμε 15 χώρες στο φόρουμ υψηλού επίπεδου και πρόκειται εκεί να αναφερθούν στο τι γίνεται σε κάθε χώρα όσον αφορά αυτούς τους στόχους του θεματολογίου 2030. Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, η Λετωνία, Λιθουανία, η Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και επίσης η Ελβετία. Πρόκειται για μια υπέροχη ευκαιρία ούτω ώστε να προσπαθήσουμε για αυτές τις κυβερνήσεις να μας λάβουν υπόψη να μας προσέξουν τώρα κάτι άλλο για το οποίο θα σας μιλήσω. Είναι το... Τώρα είναι σημαντική η υπόθεσή μας. Και έτσι να μπορέσουμε αυτού του είδους το θεματολόγιο να το συνδέσουμε με την ε, σύμβαση του ΒΕΙ για τα πρόσωπα με αναπηρία εδώ. Υπάρχει μια ομοιότητα, μια συνάφη μεταξύ των δύο μηχανισμών της προστασίας. Ε, που προβλέπονται για μας και οι δύο αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να ενσωματωθούν στην νομοθεσία, στις πολιτικές, στους προϋπολογισμούς των πατρίδων μας, ούτω ώστε κανείς να μην χάσει το τρένο και η σύμβαση του ΟΗΕ εστιάζεται στα προβλήματά μας, αλλά το ίδιο ισχύει και για το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης, οπότε και έτσι εμπλεκόμαστε άμεσα. Θα πρέπει οι οργανώσεις μας να τοποθετηθούν. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια στάση ενεργή, δυναμική και έτσι να συνδεθούν ε, αυτές οι δύο υποθέσεις και σε εθνικό επίπεδο να μας υπολογίσουν όσον αφορά την ε, εφαρμογή της σύμβασης του ΟΕΕ και την υλοποίηση των βιώσιμων στόχων και υπάρχουν κάποιες ε, μεταβλητές. Έχουμε επίσης κάποια επικάλυψη μεταξύ των δύο αυτών ε, συνθήκων, μεταξύ των δύο υποθέσεων. Και μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουμε δύο στόχους που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι άσχετοι από τη δική μας υπόθεση. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ε, ας πούμε τα οικοσυστήματα ε, που αφορούν την επικράτεια, το έδαφος, δηλαδή ότι είναι κάποια θέματα που δεν μας αφορούν. Όμως έχουμε 16 στόχους αυτού του θεματολογίου, έχουμε ένα 15-15, συγγνώμη διορθώνει, 15 στόχοι του θεματολογίου μας αφορούν και ε, αυτό αφορά τη σύμβαση του ΟΗΕ που θα πρέπει να συνδέσουμε με τους στόχους τους βιώσιμους και με τις προσπαθίες μας. Επίσης, θα πρέπει οι φορείς μας να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να μάθουμε τι γίνεται με αυτούς τους στόχους. Θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε το θεματολόγιο στο έργο μας, στη δουλειά μας. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε μια στάση δυναμική όσον αφορά αυτή την υπόθεση της ανθρώπινης ανάπτυξης και επίσης εμείς θα πρέπει να καταφέρουμε το ότι όταν οι κυβερνήσεις κάνουν το δικό τους θεματολόγιο για το θεματολόγιο 2030, ε, τότε οι κυβερνήσεις μας να μας λαμβάνουν υπόψη. Κανείς δεν θα το κάνει αντί για μας και για μας. Αν εμείς δεν μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις κυβερνήσεις μας, ε, τότε από μόνη της κάθε κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάτσει και να σκεφτεί ότι τόσο άμεσα αφορά εμάς αυτό το θεματολόγιο. Και επίσης έχουμε πάρα πολλούς τομείς, ε, πάρα πολλές, πάρα πολλούς φορείς της κοινωνίας που αφιερώνουν πόρους σε αυτή την ανάπτυξη και να εξασφαλίσουμε ότι και σε αυτονών τις προσπάθειες, όπως έλεγε ο Επίτροπος να εμπλακούμε αλλά χάρη στο έργο μας θα πρέπει παντού να φτάσει το μήνυμα γιατί οι δωρητές είμαστε και εμείς οι οργανώσεις μας άρα θα πρέπει να εμπλακούμε και εμείς οπότε θα πρέπει να υπάρξει και συνεργασία με τρίτες χώρες σύμφωνα με το θεματολόγιο αλλά και εκεί θα πρέπει να εμπλακούμε για το τι γίνεται στη χώρα τη δική μας, σε μια αδελφή χώρα, τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και έξω από αυτήν, φίλοι και φίλες, εκπρόσωποι των προσώπων με αναπηρία, να χρησιμοποιήσουμε το θεματολόγιο 2020-2030, ούτω ώστε μια τέτοια συνεργασία, μια τέτοια αμοιβαία αρρωγή μεταξύ αδελφών χωρών να μας οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου. Κανείς να μην μείνει πίσω. Αυτό πάει να πει να μείνει πίσω κανείς από μας, άντρες και γυναίκες. Ακόμα και με όσους ακόμα δεν έχουν εμπλακεί στο έργο μας. Όλοι στο αναπηρικό κίνημα, όσοι ακόμα δεν έχουν συμμετάσχει, θα πρέπει να εμπλακούν και αυτοί που δεν έχουν ορατές, αισθητές αναπηρίες. Όπως έλεγαν οι τυφλοί και κόφοι φίλοι, αυτό είναι μια καλή ευτυχή συγκυρία. Δεν θα πρέπει κανείς να μείνει πίσω και ιδίω να προσέξουμε το θέμα των αναπήρων γυναικών και ανηλίκων γυναικών. Έχουμε διάφορα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της ισότητας, αλλά αυτά τα μέτρα δεν καλύπτουν εμάς τις γυναίκες με αναπηρία, τις ανήλικες γυναίκες με αναπηρία. Πρόκειται για μία στις έξι. Άρα θα πρέπει και αυτό να καλυφθεί από την βιώσιμη ανάπτυξη, η ισότητα των φίλων. Κανείς δεν μας αφήσει απ' έξω. Many thanks, Anna. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Μα υπενθύμησε ότι έχουμε δύο ισχυρά εργαλεία στη διάθεσή μα. Έχουμε του στόχου τη βιώσιμου τη ε, ανάπτυξη, ε, την Ατζέντα ε, για το 2030 και το CRPD, την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία. Έχουμε καθυστερήσει όμω πολύ και θα να σας ευχαριστήσω καταρχάς που είστε ακόμα εδώ όσοι έχετε μείνει εδώ. Θα μετρήσουμε πραγματικά το χρόνο ομιλία. 1,5 λεπτό αντί για 2 λεπτά γιατί ιδάλλως δεν θα έχουμε καθόλου τερμηνία. Το λόγο έχει ο Μάικλ Κάμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δυσλεξία. Έχετε το λόγο. Μάικλ Κάμ, είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δυσλεξία και μιλώ για τους Ευρωπαίους που πλήττονται από μια όρατη αναπηρία. Η δυσλεξία, η δυσλεξία είναι πιο ευρέως τα δεδομένη δυσκολία, ε, εκπαιδευτική και μαθητική δυσκολία που παρεμποδίζει την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και δυσκολεύει την όλη διαδικασία και άλλες διαδικασίες. Περιλαμβάνει η ομάδα αυτή 10 έως 15% του συνολικού πληθυσμού η ικανότητα ανάγνωση και γραφής είναι σημαντικές προϋποθέσεις στις κοινωνίες μας για τα άτομα, για κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς για την επιτυχία του ατόμου. Τα άτομα με αναπηρία λοιπόν, με την δυσλεξία, ουσιαστικά πλέουν σε έναν κόσμο αρνητικό και εχθρικό προ την δυσλεξία. Αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στο σχολείο, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση. Έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τη γενική του επικοινωνία, σε ό,τι αφορά και την κοινωνική του ζωή. Επηρεάζονται προφανώ και οι ίδιοι και τα μέλη τη και όλη η κοινωνία. Εκατομμύρια λοιπόν παιδιά έφηβοι και ενήλικοι με δυσλεξία σε όλη την Ευρώπη έχουν δικαίωμα να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικέ του ευκαιρίες. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεργαστούν με την Ένωσή μας για να είναι έγκαιρη η διάγνωση περιπτώσεων δυσλεξίας στην Ευρώπη και να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση διαβίου και να καταστεί πραγματικότητα οι ίσες ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λεκή Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάρτιν Γκέικ από το Σλοβενικό Εθνικό συμβούλια, αν είναι ακόμα μέσα στην αίθουσα, έχετε το λόγο παρακαλώ. Θα I will give λοιπόν, δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, κ. Ξέντερλο, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα άτομα με αναπηρία. Εξ ονόματος του SPD θα ήθελα να δώσω τρία μηνύματα, αν με επιτρέπετε. Δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ. Αυτό το μήνυμα θεωρώ πέρασε. Χωρίς ε, την ε, συμπεριλήψη και των ε, βιώσιμων στόχων καλούμε για πολιτικό συντονισμό και θέλουμε ένα σαφή προϋπολογισμό προκειμένου αυτές οι δύο σημαντικές πολιτικές να συνενωθούν. Αλλά ας μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ EDF και κλιματικής αλλαγής. Χάρη λοιπόν στην ε, EDF και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη έχει καταστεί μια πιο συμπεριληπτική και ζεστή κοινωνία. Σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά για την 20η επέτειό σας. Δεύτερο μήνυμα να βάζουμε τα μέσα εκεί που χρειάζονται. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει υψηλά πρότυπα για τη δαπάνη των κοινωτικών πόρων, για τα διευθυντικά ταμεία. Υπάρχει όντως εξαντερετικότητα, ρεσιμότητα εκ των προτέρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα διοχετεύονται σε παροχημένα μοντέλα παροχής υπηρεσιών. Θέλουμε τα, τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρχές σε όλες ε, τις μεθόδους βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτο μήνυμα, να επενδύσουμε στον κόσμο. Δέκα χρόνια μετά την κρίση ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει μια στρατηγική κοινωνικών αποδομών, να προωθήσει την ανάπτυξη με μονομένων και ειδικών συστημάτων υποστηρίξης εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αυτά τα συστήματα δεν θα πρέπει να αποτελούν ε, απορία συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Και τα άτομα λοιπόν με αναπηρία θα πρέπει να είναι σε ηγετική θέση σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που τους αφορούν. Κλείνοντας, να πούμε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, αλλά θα πρέπει ο κόσμος μας να καταστεί πιο ζεστός και πιο ευπρόσδεκτος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Χέλγα Στίβενς, Ευρωβουλευτής. Thank you. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ε, οι 195 χώρες που κύρωσαν την ε, σύμβαση του, ΕΕ, γιατί μην ξεχνάμε ότι και πολλές άλλες χώρες διεθνώς πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυρώσει αυτή την σύμβαση του Έχουμε ένα συνασπισμό διεθνή λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ, αλλά έχουμε και την, ε, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία κάτι που υπάρχει παγκοσμίω, θα πρέπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουμε κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και θα ρίνω το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία να σκεφτεί πιθανές διεθνείς συμμαχίες. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλούμε για χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας, Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ο σημαντικότερο αναπτυξιακής αναπτυξιακή στον κόσμο. Αλλά πού Πού έχουμε την ε, διάσταση της αναπηρίας στην αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουμε. Συνεκτιμάμε και το θέμα αυτό. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε πολλές εταιρικέ σχέσεις με κοινοβούλια και άλλων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε και τη σκοπιά των ατόμων με αναπηρία σε όλες αυτές τις συνεργασίες που έχουμε με άλλα κοινοβούλια και άλλες κυβερνήσεις. Ε, Έχω πάει στο Καζακστάν, Κυριζία, Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν ως μέλος ε, της ε, αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές και σε κάθε ταξίδι τονίζω τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και πόσο σημαντικό είναι να τα λάβουμε υπόψη. Επίσης είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε τις εμπειρίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ακούμε τις δικές τους εμπειρίες και να καταλήξουμε σε κοινή ερμηνεία για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει μερικές φορές να εξηγούμε τα πιο δυσνόητα τμήματα αυτής της Σύμβασης. Αυτό το τονίζω εγώ σε όλες τις αποστολές που πραγματοποιώ στα, πλαίσια της αντιπροσωπείας στην οποία συμμετέχω. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, Σωτήρη Ξιούρο από την Κυπριακή Συνομοσπονδία των Αναπηρικών Οργανώσεων. Κύριε Πρόεδρε, επιφανείς καλεσμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την ευκαιρία που μας δίνεται να κάνουμε έστω και μια σύντομη παρέμβαση σε αυτό το τέταρτο Ευρωκοινοβούλιο των ατόμων με αναπηρίες και να σας μεταφέρω ε, τη Σκοπιά και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Αναπηρικών Οργανώσεων. Θα θέλαμε σήμερα να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ε, κέρυες ε, και κρίσιμες προπλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στις πατρίδες μας. Για παράδειγμα, η εφαρμογή της ε, διεθνούς ταξινόμησης της λειτουργικής αναπηρίας και της υγείας, καθώς και τη συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας στην ανάπτυξη πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης, θα πρέπει να διαλέξουμε ένα μοντέλο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα προσαρμόζεται στην αναπηρία και θα τηρεί και θα σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής το σύστημα ε, αξιολόγησης της λειτουργικότητας και της αναπηρίας χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ε, ετούντων στις και δικαιούχων σημαντικών επιδομάτων προκειμένου να υλοποιήσουν ένα αξιοπρεπές ποιοτικό επίπεδο και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες. Λόγω του περιορισμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και εξαιτίας του αποκλεισμού πολλών από το κράτος πρόνοιας η αδικία και ανισότητα που μαστίζει κυρίως τα άτομα με αναπηρία συνεχίζεται και αυξάνεται. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με τη βοήθεια της οικογένειας πολλά άτομα με αναπηρία είναι σε θέση να έχουν σημαντικές δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά έχουν υποστεί περικοπή των επιδομάτων τους ή έχουν στερηθεί τη, την 24ωρη προσωπική βοήθεια που χρειάζονται. Αυτή δυστυχώς είναι μια στιγμή και ταπεινωτική κατάσταση που τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να ανεχτούν. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη λήψης μέτρων από τα κράτη-μέλη με τη συνεισφορά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει την Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών και ελπίζω να τροποποιηθεί το ισχυρό σύστημα αξιολόγησης και να αντικατασταθεί από ένα καταλληλότερο μηχανισμό που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε, αλλά πρέπει να περάσουμε στον επόμενο μιλητή, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θα δώσω το λόγο στον Herbert Pichler από το Αυστριακό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία. Λυπάμαι που σας κόβω, αλλά σας θέλω παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Ο κύριος Herbert Pichler. Στο 671 κάθομαι. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είμαι σύντομο. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο σημείο 4, η κατάρτιση. Καθίσταται διαρκώ και πιο σημαντική. Αποτελεί ένα από του δικού στόχου τη Ομοσπονδιακή ε, Κυβέρνηση τη Αυστρία είναι να επανέλθουμε στο σύστημα των ειδικών σχολείων. Και αυτό πρέπει να σα πω ότι μα δυσκόλεψε ιδιαίτερα και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την αποφύτιση, την, το δίπλωμα, να ακολουθήσει κανείς σε σωστές σπουδές, σε ευρωπαϊκές σπουδές. Οι πιο πολλοί έχουν καταλήξει σε ιδρύματα που ουσιαστικά σε δουλειές που τους αποφέρουν μόνο χαρτζηλίκη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να απομακρυνθούμε αυτά τα ειδικά σχολεία να είναι κοινή η εκπαίδευση για όλους σε ό,τι αφορά και τη μετέπειτα απασχόληση, σε ό,τι αφορά την εκδήλωση. Θα ήθελα να συγχαρώ τους οργανωτές για το γεγονός ότι κατάφεραν να διοργανώσουν μια τόσο εξαιρετική συνεδρίαση με τόσους πολλούς συμμετέχοντες, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ενδεχομένως αυτή η εκδήλωση θα έπρεπε ίσως να παίρνει δύο ημέρες, γιατί βρίσκω ότι είναι πραγματικά κρίμα και άδικο να τρέχουμε τόσο πολύ. Και έτσι λοιπόν μετά από ένα λεπτό και θα σταματάω και ζήτω η Ευρώπη. Σα ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στην Σουζάνα. Τη Σουζάνα Σιλιβάνα για τον αυτισμό στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Πριν από 14 χρόνια έγινα ακτιβίστρια γιατί δεν μπορούσα να βρω σχολείο για το παιδί μου 7 χρονών τότε και υπέφερε από αυτισμό. Θεωρούσα ότι ήταν αδύνατον στον 21ο αιώνα στην Ευρώπη να υπάρχουν τέτοια προβλήματα, άρα άρχισα να μελετώ την νομοθεσία από μόνη μου για να τον υποστηρίξω. Τώρα είμαι επικεφαλή μια ε, Ευρωπαϊκή διεθνούς μάλιστα, ε, οργάνωσης και κατά πολεμό. μάλλον ω ακτιβίστρια προασπίζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών και ξέρω ότι δεν είμαι μόνη μου. Ένα στου 100 ανθρώπου ζει με αυτισμό. 7 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη και σε ορισμένε περιπτώσει έχω την εντύπωση ότι τα άτομα με αυτισμό είναι ακόμα σε πιο μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλα άτομα με αναπηρία. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν το εξή. Πόσε εθνικέ αντιπροσωπείε έχουν συμπεριλάβει άτομα με αυτισμό στους κόλπους της ομάδας. Θεωρώ ότι δεν θα είναι πολλέ αυτές οι πολιτικές ομάδες. Επίση διαπιστώνω ότι δεν είναι μόνο το παιδί μου που ζει με τον αυτισμό πολλά άλλα παιδιά είναι περιθωριοποιημένα και δεν μπορούν να συμμετάσχουν ε, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή. σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, πάνω από το 50% των παιδιών αυτών εξαιρούνται, αποκλείονται μάλλον από την εκπαίδευση αυτή. Και μια άλλη παρόμοια έρευνα καταδεικνύει ότι πάνω από το 66% των ενηλίκων με αυτισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ε, αγορά εργασίας Κλείνοντα να πω ότι είναι ωραίο και θετικό να υπάρχουν αυτά τα διεθνή έγγραφα, η σύμβαση του ΟΗΕ, οι βιώσιμοι αλλά κάτι λείπει, λείπει η εφαρμογή, η υλοποίηση και η παρακολούθηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρίνα Σουπίνα από την Διεθνή Ομοσπονδία των Νέων Βαρικών. Οι έχουν ε, μια αναπηρία που δεν είναι ορατή. Πολλές φορές ε, του, τους ξεχνούν. Ε, πολλές φορές το μεγάλο πρόβλημα είναι το πώς θα έχουν πρόσβαση σε κάποια τεχνολογία που θα τους βοηθήσει για εκπαίδευση, παιδεία, απασχόληση. Και σήμερα βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα ε, όπου υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά αυτό το σύστημα υποτιτλισμού. Πολλοί νέοι δεν έχουν δουλειά. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά ε, αν δεν έχουν κάποιο βοήθημα για την ακοή. Και δεν μπορούν να βρουν τέτοιο βοήθημα, όμως αν δεν έχουν τη δουλειά να τους δώσει τα χρήματα για να το αγοράσουν. Φαύλο κύκλο. Δεν είναι δυνατόν να πάρουν συνταγή για ένα κατάλληλο τέτοιο βοήθημα. Οπότε, το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά έχουν μια δουλειά χαμηλών δεξιοτήτων, παρά το ότι έχουν καταβάλει σκληρές προσπάθειε ε, στα πλαίσια της μόρφωσης και εκπαίδευσής τους. Μα τι γίνεται με όλα τα επιτεύγματα σε επίπεδο τεχνολογίας και αποκατάσταση των ε, προβλημάτων της υγείας. Προς τι όλα αυτά. Θα πρέπει να αναγνωστεί το δικαίωμα μας να μπορούμε να έχουμε κάποιες συσκευές που να μας ε, βοηθούν και χρειάζεται κάποιο σύστημα επιστροφών ιατρικών εξόδων. Είναι θέμα κοινωνικό, όχι μόνο ιατρικό για τους νέους. Οπότε Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι να κάνει όσον αφορά αυτά τα βοηθήματα της ακοής. Να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα επιτροφής των εξόδων. Να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο έρασμος, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα αντίστοιχα προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτά που προβλέπονται για τους νέους με αναπηρία. Τέλος, απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει πρωτοπορία όσον αφορά την υιοθεσία κάποιων ε, προτύπων όσον αφορά τα βοηθήματα ακοής, ε, τον υποτιτλισμό και τα άλλα βοηθήματα που μπορούμε να έχουμε την τεχνολογία. Σας ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στον Chris Roberts από την Alzheimer Europe ε, αν είναι ακόμη παρόν στην αίθουσα. Diagnosed My name Chris. Ονομάζομαι Chris Roberts. Διαγνώστηκα με Alzheimer πριν από πέντε χρόνια. Και Άνια. Ε, και μάλιστα εκπροσωπώ την ε, Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασία για την Άνια, που είναι ένα είδο αναπηρία, ε, που υπόκειται σε διακρίσει, σε περιθωριοποίηση. Και σε διεθνέ επίπεδο το αντίστοιχο είναι η Σύμβαση των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία, το CRPD. Ε, μιλούμε για προσαρμογές που χρειάζονται και διαρρυθμίσεις ώστε ε, όσοι έχουν άνοια και άλλες ε, αναπηρίες ε, να συμμετέχουν και να μην αποκλείονται. Θέλουμε οι υπηρεσίες που υπάρχουν να βοηθούν τη μείωση του άγχους ε, και της ταραχής, της αναστάτωσης ε, των πασχόντων από άνοια. Αναστάτωση που τη βιώνουν και άγχος που βιώνουν καθημερινά και να μην ξεχνούμε και τις οικογένειες που επηρεάζονται. Επίσης, ένα τέταρτο των τροφίμων φυλακών και νοσοκομείων έχουν άνοια. Πώς θα διευκολύνουμε τη δική τους καθημερινότητα και δυστυχώς καλές πρακτικές ε, δεν είναι αρκετά διαδεδομένες. Ε, χρειάζεται κατάρτιση, χρειάζεται συνειδητοποίηση του προβλήματος για να βελτιώσουμε αυτή, ε, αυτό το σύστημα που είναι ατελές. Και όσοι πάσχουν από άνοια αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και στιγματίζονται, είναι θύματα προκαταλήψεων. Δεν υπάρχει ακόμη κατανόηση για την ασθένεια αυτή. Και είναι τόσο πολλαπλές οι διακρίσεις ε, που προστίθεται στις διακρίσεις λόγω ηλικίας ή ε, φύλου. Ε, υπόκειται σε επανοχλήσεις, υφίστανται την ε, έλλειψη υπηρεσιών και δυστυχώς δεν υπάρχουν φορείς που να μας προστατεύουν. Είναι πολύ διαφοροποιημένη η μεταχείριση και σε μερικές περιπτώσεις αγνοούνται τελείως τα δικαιώματά μας. Και πολλοί πάσχοντες από άγνοια δεν γνωρίζουν τους νόμους που υποτίθεται ότι πρέπει να τους προστατεύσουν. Ε, μάλιστα μερικές φορές επειδή η άνοια είναι αόρατη, ε, πολλοί κόσμοι την αγνοεί. Ε, και οι ανάγκες των πασχόντων που είναι πολύ διαφορετικές ανάλογα με το πόσο προχωρημένο στάδιο είναι το περιβάλλον του την ηλικία του, την υποστήριξη που λαμβάνουν, την έλλειψη υποστήριξης που εκείλουν ε, οι ανάγκες. Γι' αυτό το μοντέλο αναπηρία ε, που ε, κανονικά θα έπρεπε να εφαρμοστεί για την άνοια παραγωνίζεται. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ όσους παρέμειναν για να ακούσουν, για να μην αφήσουν ούτε εμάς πίσω. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. I will give the floor now to A.B. Akram for one minute, if you can, please. Thank you very Το λόγο έχει Άμπι Άκραμ για ένα λεπτό. Εκ μέρους ε, των, ε, της ομάδας ε, γυναικών με αναπηρία από όλο τον κόσμο θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε ουσιαστικά το σύνθημα να μην αφήσουμε κανέναν πίσω θα τα καταφέρουμε μόνο αν συμπεριλάβουμε και τις γυναίκες με αναπηρία ε, στις ηγετικές θέσεις. Για... Μόνο έτσι θα πραγματώσουμε το σύνθημα να μην μείνει κανένας πίσω. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ικανότητες των γυναικών και το πώς αντιλαμβάνονται το σώμα τους, τα δικαιώματά τους. Πολλές είναι οι, οι γυναίκες με α, με αναπηρία και οικογένειες, ε, πολλές φορές οι οικογένειές τους τις ε, θεωρούν βάρος. Και ελάχιστε είναι οι εκπρόσωποι των γυναικών με αναπηρία στις οργανώσεις. Πώς θα γεφυρώσουμε αυτό το κενό. Θα πρέπει η πολιτική ε, και η θεσμική συνοχή να βελτιωθούν. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την ηγετική ικανότητα και των γυναικών. Μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε τις αλλαγές με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα με συμμετοχή σε κάθε χώρα, αλλά και περιφερειακούς μηχανισμούς ε, ενσωμάτωσης των γυναικών. Ευχαριστώ. Really but now... που ε, από το χρόνο αλλά τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο για να κλείσουμε και λυπάμαι ιδιαίτερα, αλλά είχαμε καθυστέρηση προηγουμένως. Colleagues, uh, Συνάδελφοι, ε, φίλοι, πριν πω δύο λόγια για να κλείσουμε αυτή την πολύ επιτυχημένη ε, εκδήλωση. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Νότον που δούλεψε άκοπα μέρες ολόκληρες με την ομάδα του για να καταστήσει δυνατή αυτή την ε, εκδήλωση. Κάρστον, λοιπόν, ε, θα ήθελα να πεις δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι ιδιαίτερα... Έχω αντίληψη ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ήθελαν να πάρουν το λόγο και δεν μίλησαν. Αν είσαστε στον κατάλογο των ομιλητών και δεν καταφέρατε να πάρετε το λόγο σας, παρακαλώ στείλτε την παρέμβασή σας για να τη δημοσιεύσουμε. Για να μπορέσουν όλοι να τη διαβάσουν. Σας παρακαλώ λοιπόν στείλτε τι μας και Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη από τη δουλειά που κάνατε όλοι σας. Από τη δουλειά που έχουν κάνει και οι βουλευτές και από όλη την κινητοποίηση που υπήρξε. Εκτίμησα πραγματικά όλες σας τις παρεμβάσεις, όλες σας τη δουλειά σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Αγαπητά μέλη. Η σημερινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχη. Το γεγονό. ότι έχουμε περίπου 800 εκπρόσωπους οργανώσεων ατόμων με αναπηρία από όλη την Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη. Το ότι ήρθατε να συμμετάσχετε στη σημερινή εκδήλωση το γεγονό αυτό καταδεικνύει ότι το κίνημα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη είναι πιο ισχυρό παραποτέ. Επίσης όμως η περίοδος στην οποία διανύουμε είναι και πιο δύσκολη από ότι οι προηγούμενες και θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Για μας λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, η σωστή ισορροπία σημαίνει ακούραστη εργασία για τη βελτίωση των οργανώσεών μας προκειμένου να, προκειμένου να τις καταστήσουμε πιο συμπεριληπτικές, προκειμένου να έχουν πιο πολλά μέλη για να δημιουργηθεί χώρος, πιο πολύς χώρος για τα μέλη αυτά των οργανώσεών μας που πλήττονται πιο πολύ από όλους για να ακουστούμε με τους αριθμούς μας, με την αριθμητική ισχύ μας. Δεν αρκεί να λέμε ότι α, εκπροσωπούμε 80 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε αυτόν τον αριθμό να λειτουργήσει υπέρ μας. Και αυτό πώς θα το πετύχουμε. Πρέπει να κάνουμε αυτά που συμφωνήσαμε, τι συμφωνήσαμε. Καταρχάς, για το μανιφέστο, συμφωνήσαμε επί του μανιφέστου για τις ευρωεκλογέ. Αφότου το εγκρίναμε, συμφωνήσαμε να ξεκινήσει η εκστρατεία. Η εκστρατεία θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα το 2019 να ψηφίσουν πιο πολύ στις ευρωεκλογέ, να έχουν εκλογικό δικαίωμα, δικαίωμα ψήφου πιο πολλά άτομα με αναπηρία στα κράτη-μέλη και να εκλεχθούν και πιο πολλά μέλη με αναπηρία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή η εκστρατεία λοιπόν θα πρέπει να προωθηθεί από όλους μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ε, συμφωνήσαμε να ξεκινήσει και μια δεύτερη εκστρατεία για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2020 μέχρι το 2030. Συμφωνήσαμε λοιπόν επί του ψηφίσματος, το ψηφίσαμε, το εγκρίναμε Χρειάζεται υποστήριξη από τις πρωτεύουσε. Και η δουλειά αυτή θα γίνει και στις Βρυξέλλες, χέρι-χέρι. Και επίσης, πριν από αυτό, συμφωνήσαμε επίσης η Ευρώπη να αποτελεί παγκόσμια ηγέτητα σε ό,τι αφορά την πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Την ε, υπερληπτική ανάπτυξη, την εφαρμογή των στόχων των βιώσιμων της βιώσιμης ανάπτυξης με καθοδήγηση από τη συνθήκη, τη σύμβαση του ΟΕΑ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ούτω καθεξής. Άρα όλα αυτά τα οποία συμφωνήσαμε θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην καθημερινή μας ατζέντα. Ακόμα και αν προερχόμαστε από μια οργάνωση από ένα μικρό χωριό θα πρέπει να τα εντάξουμε όλα αυτά στην καθημερινότητά μας, στην δική μας ατζέντα. Αν στη μελλοντική σας, ε, στο μελλοντικό σας δρόμο διαπιστώσετε ότι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία δεν κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνει, τουλάχιστον να κρούσετε τον κόδωνα. Και εμείς θα, θα σας εισακούσουμε. Τουλάχιστον όμως να χτυπήσετε το κουδούνι. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αμοιβαιότητα, είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση και εμείς θα σας κρούσουμε τον κόδωνα. Τώρα, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περαιτέρω και να σας απασχολήσω άλλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Επιτρόπο, τον Πρόεδρο Ταγιάννη για τη δέσμευσή του, για την υποστήριξή του, για την συμμετοχή του την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του και όχι μόνο για τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και για άλλα στοιχεία. Να ευχαριστήσω επίση τα μέλη τη διακομματική ομάδα για τα άτομα με αναπηρία για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει ω τώρα και που αναμφίβολα θα συνεχίσουν στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου επίση που σα υποστήριξαν και εσά και άλλου και μπορέσατε να βρίσκεστε εδώ σήμερα. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου όλους όσοι εργάστηκαν αποτελεσματικά, αποδοτικά με την Κάρσταν και με το προσωπικό μας προκειμένου να καταστεί δυνατή η σημερινή εκδήλωση. Πριν από κάποια ώρα, ένα συνάδελφο είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαζόμασταν δύο ημέρε. Αυτό ενδεχομένω να το εξετάσουμε ω προοπτική για το μέλλον. Νομίζω πως οι βουλευτέ θα μπορούσαν να φροντίσουν για μία ακόμα ημέρα. Θα υπήρχε μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Θα μας επέτρεπε αυτό να δουλέψουμε και σε υποεπιτροπές, να συζητήσουμε πιο πολλά πράγματα, γιατί υπάρχουν πραγματικά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και χειρό. Θα γυρίσουμε πίσω, θα επιστρέψουμε. Έχουμε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες. Αυτή η εκδήλωση να λαμβάνει χώρα μία φορά σε κάθε θητεία του Κοινοβουλίου. Η πέμπτη λοιπόν θα λάβει χώρα μεταξύ του 2019 και του 2024. Να ευχαριστήσω επίσης τους Δερμηνείς, όλους τους Δερμηνείς. Πολύ Που ε, κατέστησαν δυνατή την επικοινωνία και αποτελεσματική μάλιστα. Και εμεί σα ευχαριστούμε και προφανώς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, τον καθέναν από εσά που είσαστε εδώ σήμερα. Σας παρακαλώ να μεταβιβάσετε το μήνυμα αυτό στις πατρίδες σας, γιατί το σύνθημα «Τίποτα για μας χωρίς εμάς» συνεπάγεται ένα τρόπο διοργάνωσης του διαλόγου, συνεπάγεται ένα τρόπο διοργάνωσης της ίδιας της δημοκρατικής διαδικασίας και να είστε ε, ευγενείς σε όσους σέβονται την αρχή αυτή και σκληροί σε όσους δεν τη σέβονται για τη τελική ανάλυση. Όταν κάποιος ε, είπε ότι είμαστε πολύ ενθουσιώδεις και είμαστε με στο χαμόγελο εδώ, ε, εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι ναι, αλλά είμαστε και εξίσου αποφασισμένοι. Είμαστε αποφασισμένοι και να είστε αποφασισμένοι να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας. Σας ευχαριστώ όλους. Thank you for taking over and choosing the meeting. Didn't give me the paper. Give me please that I can say the flight. Υπότιτλοι AUTHORWAVE